Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε και στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα έχουμε μέχρι τις 3.30 μια δημόσια κρόαση. Θέμα αυτής θα είναι η εποχή μετά την Αραβική Άνοιξη και η πορεία στη περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Μετά τι εξηγήσει του 2011, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ την κατάσταση στην περιοχή. Είχαμε μάλιστα πολύ άριθμε ανταλλαγέ απόψεων και πολλέ ε, αποστολέ στι χώρε ΜΑΒΑ. Και πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στην αίθουσα συμμετείχαν ενεργά σε αυτέ τι αποστολέ. Και είναι πολύ έγκαιρη και επίκαιρη αυτή η έκθεση ώστε να κάνουμε ένα απολογισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή αυτή και να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε και την αποτελεσματικότητά της. Επίσης, χάρη στην έκθεση αυτή και στο τέλος της κοινοβουλευτικής αιτίας θα αξιολογήσουμε ποια είναι τα μέτρα στήριξη ε, προ χώρε αυτέ ε, και τι πρόθεση των δημοκρατικών του βλέψεων και θα δούμε που, σε ποιους τομείς θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή μα για αυτή την έκθεση για την εποχή μετά την Αραβική Άνοιξη, τον κύριο Μπενιφέη. Σωστά κάθεστε, αλλού σα έβλεπα συνήθω. Εν πάση περιπτώσει, πριν δώσω το λόγο στον Μπράντον Μπενιφέη, τον εισηγητή μα να καλέσω του δύο καλεσμένου μα, ξεκινώντα μια αλφαβητική σειρά από τον κύριο Ούτασα Αντάμ από την Οξφάμ και Διευθυντή για το Τμήμα της Συρίας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και να καλωσορίσω θερμότητα και την Νάταλη Τότσι, τη γνωρίζουμε πολύ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών ε, Υποθέσεων και ε, σύμβουλος της ΥΠΑ της εκπροσώπου της κυρίας Μαγκερίνη. Επίσης είναι επίτιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν. Και μάλιστα γνωρίζουμε την κυρία Τότσι γιατί συνέβαλε στην διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής που περιλημμένω συζητούμε στην Επιτροπή. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπενιφέη, τον εισηγητή μας, κατόπιν στην κυρία Τότση και στο τέλος στον κύριο Μουτάς Αντάμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα και ως εισηγητή σήμερα για την έκθεση για την περίοδο μετά την, την Αραβική Άνοιξη. ορίζω και την κυρία Τότσι από το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων ε, και τον κύριο Ντάντι για την Oxfam την κυρία Ντάντι για την Oxfam ε, στο θέμα της Συρίας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν για θέμα, με θέματα μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της πολιτικής γειτονίας. Χώρες της περιοχής που τα τελευταία 8 χρόνια έχουν αντιμετωπίσει ανατροπές τεράστιες μετά την Αραβική Άνοιξη όπως ονομάζεται που προκύπτει κατόπιν ε, ως εκδήλωση μιας δυσφορίας κοινωνικής ε, για τα προβλήματα που πολλά χρόνια ε, συνεχίζονταν και που μετετράπησε ορισμένες περιπτώσεις όπως τη Συρία σε μια σύγκρουση. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να ρίξουμε ένα κοινό βλέμμα στις δράσεις της Ένωσης αυτά τα χρόνια για να καταγράψουμε που έχουμε επιτυχίες, που έχουμε επιδείξει καλές πρακτικές και που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Βεβαίως η συζήτηση θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε περαιτέρω στα θέματα αυτά για να προχωρήσει η δουλειά μας στην έκθεση. Η Ένωση στις Αραβικές Ανοίξεις ε, καταρχάς αντέδρασε ε, ενθαρρύνοντας τα, τα μαζικά κινήματα στη δεκαετία του, στο, κατά τη διάρκεια του 2011. Μετά όμως με την ανάδειξη της τρομοκρατίας, του ΙΣΙΣ και του ΙΣ μεταναστευτικής κρίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε περισσότερο στην ε, ασφάλεια, τη σταθερότητα των κρατών αυτών και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Μια νέα πολιτική λοιπόν γειτονίας για το 2015 με την έκθεση ε, και την καταγραφή των καταστάσεων εκδόθηκε που εκδόθηκε και επίσης έχουμε την έννοια της, ε, του co-ownership με τους ε, στόχους και τις προτεραιότητες που συμπροσδιορίζονται με τις χώρες εταίρους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό μπορεί να θεωρήθηκε ότι το επιβάλλει άνωθεν ε, και προς τους αποδέκτες αυτής της πολιτικής. Βεβαίως η Ένωση αναγνωρίζει ότι η επίδραση της επιρροής στην περιοχή αυτή είναι περιορισμένη και βεβαίως αυτό μπορεί να είναι σωστό παρότι δεν μπορούμε να απαρνηθούμε τις αξίες μας και στις ε, χώρες αυτές και σε σχέση με τις χώρες αυτές. Ύστερα από δύο χρόνια λοιπόν υλοποίηση αυτής της νέας πολιτικής γειτονίας βλέπουμε ότι αυτές οι πολλές φορές αυταρχικές κυβερνήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και την ασφάλεια σαν να ήταν ένα αντάλλαγμα επιτρέψτε μου τον όρο έναντι της ε, του κλεισίματος του ματιού τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ανθρωπιστικής προστασίας και των ανθρωπινών δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου. Εδώ με το co-ownership έχουμε μια έννοια διαφοροποίηση, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποιες κοινέ τάσει, ωστόσο στις περιοχές αυτές, μόνο που η ιστορία, οι ιστορικές καταβολές αλλά και οι οικονομικές εξελίξεις αλλά και η έκβαση των γεγονότων που ξεκίνησαν το 2011 είναι πολύ διαφορετικές και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα προσδορίσουμε μια αποτελεσματική δράση. Ε, η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης προχώρησε με την ε, παγκόσμια στρατηγική του 2016 για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών σε διάφορους κλειδονισμούς σταθερότητα λοιπόν που αφορά τόσο κράτη όσο και οι κοινωνίες. Και είναι πολύ σημαντική έννοια, με, καθώς αλλάζει προσέγγιση, πρόκειται για μια αλλαγή υποδείγματος για τις κοινωνίες της και την κοινωνία των πολιτών που αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο ως παράγον αλλαγής και ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε τη στρατηγική προσεκτικά βλέπουμε ότι ένα κράτος ανθεκτικό είναι αυτό στο οποίο έχει ανθεκτικότητα και η ίδια η κοινωνία με τη δημοκρατία, με την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια μακροπρόθεσμη ε, σταθερότητα για τους πολίτες και ε, αυτή πρέπει να είναι και η δική μας η Το κλειδί λοιπόν για να προσαρμόσουμε τις δικές μας ε, τις ιδέες και τις προτάσεις θα είναι να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ανθεκτικότητας του κράτους και αυτής της κοινωνίας που δεν πάνε πάντα παράλληλα, κυρίως όταν πρόκειται για κράτη αυταρχικά ή ολοκληρωτικά. Ε, τα κράτη αποδέκτες επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπό το πρίσμα των προσδοκιών των πολιτών τους. Κρίση εμπιστοσύνης είναι αυτή που χαρακτηρίζει τα κράτη αυτά. Κρίση δηλαδή εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των θεσμών των κρατών αυτών και σε αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εξελίξεις. βραχυπρόθεσμα βεβαίω με λύματα όπως η ασφάλεια, η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση της μετανάστευσης είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και με τη σταθεροποίηση και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, δάλλως θα χάσουμε τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. επίση χρειάζεται μια ενότητα δράση μεταξύ των κρατών μελών, γιατί βλέπουμε ότι πολύ συχνά ε, προβάλλονται περισσότερο εθνικά, στενά εθνικά συμφέροντα και έτσι κάποια κράτη δρούν αντίθετα με τις ε, προσδοκίες ή τις επιθυμίες των άλλων κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν μια ενωμένη συνεκτική πολιτική. Η Νάταλη Τότσι θα μπορούσε νομίζω να μας πει πολλά περισσότερα για τις πτυχές αυτές και τις εκτιμήσεις της σε σχέση με την παγκόσμια στρατηγική και τα δύο χρόνια υλοποίηση τη ιδιαίτερο χαίρομαι που βλέπω εδώ που είναι, ότι είναι και η κυρία Ντάμ ε, που θα μας μιλήσει για την περιοχή αυτή γενικότερα και όχι μόνο για τη σύγκρουση στη Συρία. Μετά την ε, ενεργοποίηση αυτής της σύγκρουσης με τόσους πολλούς εταίρους, και επίκεντρο βέβαια το καθεστώς του Άσαντα έχει καθοριστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση της κρίσης με ρόλο μάλιστα ακόμη πιο λεπτό καθώς ανακοινώνεται η αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή, η ανθρωπιστική δράση την οποία έχουμε θέσει στην πρώτη γραμμή της δράσης μας με τους παγκόσμιους ε, και διεθνείς ε, παράγοντες για το θέμα των εκτοπιστέντων, των ε, μεταναστών, της υποδοχής τους στις γειτονικές χώρες αλλά και την περάτωση της σύγκρουσης. Είναι πολλές οι ανάγκες, η εκπαίδευση παραδείγματι στους τόσους νέους και τα παιδιά που έχουν χάσει τις αιστείες τους και σε αυτό θέλουμε η Όσκουσφα να, να μας πει πώς βλέπει και πώς αξιολογεί τα προβλήματα. Ευχαριστώ και πάλι τους, τις ομιλήτριες γιατί πιστεύω ή τους ομιλητές μας γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις τους για τη συνέχεια που θα δώσουμε με την έκθεση και τις δραστηριότητε της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Μπενιφέη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τότσι, την πρώτη από τους δύο καλεσμένους μας και μετά στον κύριο Μουτά Ζαντάμ. Δέκα λεπτά ο καθένας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά νιώθω που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Και η έκθεση σας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή μετά την Αραβική Άνοιξη δίνει την ευκαιρία ε, να κάνουμε ένα προβληματισμό για τις ε, πραγματικά ρηξικέλευτες ε, κοσμογονικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στην περιοχή και πώς θα προσεγγίσουμε όλα αυτά που συνέβησαν στην περιοχή Μέση Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Καταρχήν θα ήθελα να ε, επισημάνω τα τρία κατά τη γνώμη βασικά σημεία της περίοδου 2011 μέχρι σήμερα. Πρώτο θέμα, ήταν μη βιώσιμα τα καθεστώτα στην περιοχή Μάβα. Εξού και η ανατροπή τους, που είναι θέμα του πότε θα γίνει και όχι αν, κατά πόσο θα γίνει. Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο, αυτό θα ήθελα πρώτα να συγκρατήσουμε. Και το 2011-2012 κάτι τέτοιο ίσως ήταν σχετικά αναντήρητο. Το 2017 με 2018 άρχισε να γίνεται και πάλι θέμα υποσυζήτηση, να αμφισβητείτε. Φαίνεται λοιπόν ότι ξαναπέφτουμε ε, στον πειρασμό να πούμε ότι μια αυταρχική σταθερότητα μπορεί να έχει μια βιωσιμότητα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το 2011, γιατί η περίοδος τότε μας είχε αποδείξει ότι δεν ήταν θέμα του κατά πόσο, αλλά το πότε θα ανατραπούν αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Και αυτό συνέβη για κάτι που ανέφερε και ο κύριος Μπενιφέη. Το κοινωνικό συμβόλαιο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής ε, ε, καταγγέλθηκε, διεράγει και το κοινωνικό συμβόλαιο στην περιοχή αυτή έλεγε ουσιαστικά εδώ είμαστε, κυρίως αραβικά καθεστώτα που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες στον πληθυσμό σε ανταλλαγή με τη συγκατάθεση του πληθυσμού να παραμείνουν στην εξουσία. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και οι δεκαετίες, αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες δεν πια, δεν προσφέρονταν πια για πολλούς και διάφορους λόγους. Εξού και το θέμα της ανισότητας, ε, της περιθωριοποίησης που δημιουργήθηκε, ε, υπήρχε το πρόβλημα της διαφθοράς, υπήρξε και μια πραγματική έκρηξη, κυριολεκτική έκρηξη του άτυπου τομέα της οικονομίας και σε τελική ανάλυση ε, εξαλήθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στη στέγαση και στην υγειονομική περίθαλψη και ιατρική περίθαλψη. Δεύτερο κρατούμενο από την κατάσταση. Ε, αλλαγές συμβαίνουν. Αυτό φάνηκε. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Όχι, δεν είναι το θέμα πότε, αλλά αν. όχι, αν, αλλά πότε. Και μάλιστα δεν ήταν απλές αλλαγές, αλλά πολυσύνθετες και όχι μόνο περίπλοκες. Γιατί κάτι περίπλοκο συνήθως μεταξελίσσεται σε κάτι δυσδιάστατο. Αλλά κάτι που είναι πολύ σύνθετο, πολύ διάστατο, ε, φέρνει αλλαγές σε διάφορα επίπεδα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εξού και το συμπέρασμα ότι γνωρίζουμε ότι θα γίνουν οι αλλαγές, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς και με ποιον τρόπο θα συντελεστούν. Και αν εξετάσουμε τι συνέβη στην περιοχή Μέση Ανατολής και Βόρεια Αφρική από το 2011 μέχρι σήμερα, διαπιστώνουμε πως οι αλλαγέ αυτές έλαβαν χώρε σε διάφορες χώρες με διαμετρικά αντίθετου τρόπους. Είχαμε μια θετική περίπτωση όπως τη Τινησίας. Είχαμε περιπτώσεις όπου είχαμε πραγματικά μια απεγνωσμένη και άρα μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα κατάσταση, αλλά προσωρινά εμφανώς σταθερή προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από κάποια καθεστώτα που λέει δεν σας προσφέρουμε δημόσια υπηρεσία για τη συγκατάθεσή μας, σας προσφέρουμε ασφάλεια για τη συγκατάθεσή σας, για να συνενέσετε στην παραμονή μας στην εξουσία. Οπότε αυτό δεν συνιστά πρόοδο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, αλλά μια παλιδρόμηση, γιατί έχουμε μια περιχαράκωση σε απολυταρχικά καθεστώτα. Βλέπε Αίγυπτος. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου έχουμε μια κατάρρευση της κατάστασης στην Ιεμένη, τη Λιβύη, τη Συρία. Επίσης, ειδικά για τη Συρία, εκεί έχουμε πραγματικά το φίνικα, το πουλί που αναγεννάται από τις τάχτες του, αλλά δεν είναι το, ο που ξέραμε παλιά, είναι κάπως ξεποπουλιασμένος ο Φίνικας όπως έχει αναδειχθεί, αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Επίσης έχουμε αυτά τα δύο φαινόμενα που λαμβάνουν ε, παράλληλα χώρα. Από τη μια έχουμε όλο και περισσότερο χώρο περιορισμένης κρατικότητας όπως θα έλεγα και αυτή η περιορισμένη κρατικότητα παρατηρείται όχι γιατί το κράτος δεν μπορεί πια να εξασφαλίσει γεωγραφικό έλεγχο στο σύνολο της επικράτειας, αλλά είναι και ανίκανο το κράτος να ανταπεξέλθει στις βασικές του λειτουργίες. Οπότε και λειτουργικά είναι περιορισμένη αυτή η κρατικότητα. Και επίσης αυτή η ε, απίσκανση του κράτους οδηγεί σε μία μεγαλύτερη αμφισβήτηση και εκεί η συνολικότερη περιοχή ε, λαμβάνει, έχει, παίρνει κάποιο ρόλο. Γιατί στη Συρία και στην Ιεμένη είχαμε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση, ακριβώς γιατί άρχισε να γίνεται μια απονέκρωση του κράτους ή μια ένα του κράτους, της κρατικότητας. Επίσης, αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για μας τους Ευρωπαίους. Ένα σημείο που πολύ εύστοχα επισημαίνεται στην έκθεσή σας είναι η έννοια της περιορισμένης μόχλευσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλούμε για τεκτονικές ε, μεταλλάξεις που έχουν γίνει και τεκτονικούς κραδασμούς. Δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός παράγοντας που να έχει δυνατότητα επιρροής της μορφής, της μελλοντικής μορφής της ευρύτερης περιοχής ΜΑΒΑ. Οπότε δεν την έχουμε ούτε εμείς αυτή την ικανότητα ε, να ασκήσουμε τέτοια επιρροή, ούτε κανείς άλλος παγκοσμίω. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιλεκτικοί στα θέματα που διαλέγουμε. Και σίγουρα θα θέλαμε ε, μεγαλύτερη επιρροή στο Μαγκρέφ σε σχέση με το Μασρέκ. Επίσης περισσότερη επιρροή στην κατανάλωση ορεικτών καυσίμων σε σχέση με την παραγωγή, με τα κράτη παραγωγής καυσίμων. Επίσης υπάρχει το θέμα των μεγάλων και των μικρών κρατών στην περιοχή. Οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε και γεωγραφικά συγκεκριμένες περιπτώσεις και προσεκτικά. Αλλά ίσως και θεματικά θα πρέπει να επιλέξουμε που θα θέλαμε να επικεντρωθούμε. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση στην έκθεσή σας που εστιάζεται στην νεολαία και στην ιδέα ενός προγράμματος Έρασμος για την περιοχή Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Και μάλιστα και στο Ινστιτούτο μας ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά που θα βοηθήσει πολλούς νέους και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα σημαίνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Άλλο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ιδέα της ανάγκης να επικεντρωθούμε τοπικά σε συγκεκριμένα πράγματα για να έχουμε καλύτερη αντίληψη της κατάστασης. Και υπάρχει και μια άλλη πρόταση στην έκθεση που με βρίσκει σύμφωνη. Η ιδέα ότι τα γραφεία, οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να, να στείλουν ε, Συμβουλευτικέ επιτροπέ, συμβουλευτικού φορεί. και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια πιο τοπική αντίληψη του τι συμβαίνει στα συγκεκριμένα σημεία, στους συγκεκριμένους τόπους και τέτοιε αλλαγές θα μπορούσαμε να επιφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι αλλαγές Μικρή εμβέλεια δεν θα επηρεάσουν το σύνολο μια χώρας, αλλά σε τοπικό επίπεδο θα προσφέρουν τα μάλα τέτοιες αλλαγές. Ακόμη και σε εξαιρετικά περίπλοκες καταστάσεις όπως αυτές της Συρία. Εκεί βέβαια δεν είχαμε ποτέ την ικανότητα ω Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσουμε το συνολικό σχήμα που θα έχει η Σύρια στο μέλλον τη μορφή, αλλά σε τοπικό, πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ θετικό αντίκτυπο και να βοηθήσουμε στην πρόοδο. Ένα άλλο θέμα που ίσως θα πρέπει να το σκεφτείτε προσεκτικά είναι αυτή η διάκριση μεταξύ των λόγων και των έργων. Και θα σταθώ εδώ σε δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά το γενικό κοινό σφαιρικό σχέδιο δράσης και το δεύτερο είναι η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε εκπέμψει ένα χειρό μήνυμα και διατρανώσαμε τη θέση μας σε επίπεδο λόγων, αλλά τα έργα δεν ακολούθησαν. Ειδικά στο κοινό σχέδιο ε, δράσης, το σφαιρικό. Στην περίπτωση αυτή υπήρχε πρόβλημα. Γιατί και αφήνω την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Αλλά για το σφαιρικό σχέδιο διατυμπανίζαμε την αποφασιστικότητά μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προωθήσουμε όσο γίνεται το κοινό αυτό σχέδιο, αλλά όταν έφτασε ε, το χτένι στον κόμπο, δυστυχώς κολλήσαμε και δεν περάσαμε στα έργα. Και μερικές ε, φορές θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε και το τίμημα, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας. Και η περιπτώσει αυτού του σφαιρικού σχεδίου δράσης και του μηχανισμού ειδικού σκοπού ήταν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της αναντιστοιχία μεταξύ λόγων και έργων. Επίσης, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να δρούμε, όπως λέτε στην έκθεση, ως δημοκρατική ε, νομοθετική, κανονιστική, ηθική, ποιο είναι το σημείο αφετηρίας μας είναι να σεβόμαστε και εσωτερικά αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις ή ηθικές αρχές. Γιατί αν άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, ε, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Και κοιτάξτε το θέμα των μεταναστών και του ασύλου. Και αυτό δεν είναι κάτι εσωτερικό μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα του κόσμου, είναι, τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω μας. Δεν μπορούμε να λέμε ωραία λόγια και να προβάλλουμε ιδεώδη αν δεν τα τηρούμε και εμείς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τότσι. Ο κύριος Ανταμουτάζ για 10 λεπτά επίσης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίδετε την ευκαιρία να είμαι παρόν και να σας μιλήσω αυτή την τόσο σημαντική στιγμή το μέλλον και της Συρίας και της όλης περιοχής. Ο ρόλος σας είναι σφαιρικά πολύ σημαντικός και η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί και όσον αφορά τις μελλοντικές δεσμεύσεις σας στην περιοχή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να χειριστείτε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε εμείς. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για την κατάσταση στη Συρία, όπου ζω, εργάζομαι και από την ε, αρχή της κρίσης ε, ασχολούμαι με τον τρόπο με τον οποίο θα την δράσουμε στα πλαίσια της Oxford. Πρέπει να πω ότι έχουμε περίπου με ένα, πολλά προγράμματα για την παιδεία, σχέδια, για την εκπαίδευση, για το νερό, για άλλα θέματα. Μα ασχολούμεθα με υπαίθρες περιοχές ε, ε, νοτίως της Δαμασκού, στο Χαλέπη, Ανατολικά και στον Βορρά, σε όλες αυτές τις γεωγραφικές περιοχές. Κάποια από αυτά τα προγράμματα και τα project πρέπει να πω ότι χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να τα ευχαριστήσω για την υποστήριξή της. Η πρόσβαση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η πρόκληση για όποιους εργάζονται Το 2018 άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Ίσως η ΜΚΟ και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πιο εύκολη πρόσβαση. Μπορούν κάποιες ε, να έχουν ευκολότερα πρόσβαση, αλλά η πρόσβαση πρέπει να σας πω ότι γίνεται χωρίς τακτικό τρόπο. Επίσης η βιωσιμότητα του κάνουμε για μας είναι ένα μεγάλη πρόκληση, παρά το γεγονός ότι όξο και άλλες οργανώσεις μπορούν σε τακτά διαστήματα να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις κοινότητες που θέλουμε να φτάσουμε. Ποιες είναι οι άλλες προκλήσεις που έχουν σχέση με την ανταπόκρισή μας στο πρόβλημα της Συρίας. Είναι ότι έχουμε περιορισμένη χρηματοδότηση ή μη χρηματοδότηση. Δεν έχουμε αρκετά κονδύλια. Κυρίως όσοι ε, να έχονται στην περιοχή των Χαμς της Δαμασκού, όποιοι εργάζονται στα πλαίσια των κινητικών οργανώσεων ξέρουμε ότι τα δύο τρίτα των ατόμων στα οποία στοχεύουμε ζουν σε αυτές τις περιοχές. Η έλλειψη χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο μειώνει την δυνατότητά μας να ενεργήσουμε παρά το γεγονός ότι είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και την δυνατότητά μας να αναπτύξουμε περισσότερα προγράμματα και να προγραμματίσουμε. Άπιο άλλη πρόκληση επίσης είναι το ότι έχουμε κυρώσεις ε, για κάποια ε, θέματα που δημιουργούνται και δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν κονδύλια και από το εξωτερικό. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα. Προσπαθούμε στα πλαίσια της Oxfam να προσπαθούμε να πάμε στην περιοχή του Ιλτίβ. Ξέρουμε όμως ότι είχαμε προβλήματα και χρειάστηκε να σταματήσουμε. Κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσω επίσης για τη Συρία είναι ότι είναι πολύ διαφορετική από άλλες ε, χώρες της περιοχής. Σε κάθε χώρα έχουμε ένα μοναδικό μοντέλο. Στις περισσότερες αυτή οι οποίοι διαμαρτύρονται έχουν μια ελπίδα ότι στο τέλος θα υπάρξει αλλαγή. Εμείς είδαμε αλλαγές στις κυβερνήσεις, παρά το γεγονό ότι οι ελπίδες ποτέ ίσως δεν πραγματοποιήθηκαν. Στην περίπτωση όμως της Συρίας, πρέπει να πω ότι τέτοιου είδους ελπίδες πνίγηκαν αμέσως και επικρατεί μάλλον ένα στρατιωτικό κλίμα και μεγάλη αυστηρότητα. Και σιγά σιγά καταλήξαμε σε μία εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων που είναι παρούσε στη Συρία. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση σας θα πρέπει σε σχέση με τη Συρία να είναι διαφορετική από αυτή για τις άλλες χώρες, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στη Συρία. Η έκθεση για την ε, ισότητα δύο φίλου στα πλαίσια τη άνοιξη των ευρωπαϊκών οργανισμών, πρέπει να πω ότι μπορεί να περιοριστεί σε δύο γραμμέ, λέγοντα ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπογραμμιστούν στην έκθεση και θα πρέπει να αποτελέσουν και το ε, κύριο θέμα στο οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε. Κυρίω όσον αφορά τη γυναίκα. Οι γυναίκε και τα νέα κορίτσια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση παντού, να μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα προβλήματα και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να υποστηρίζονται από οργανώσεις και οι οργανώσεις αυτές να υποστηρίζουν τα προγράμματα της, του Ισόκραν στη Συρία. Πρέπει να πω ότι προσπαθεί στα πλαίσια της ισότητας των φίλων να κάνει τέτοιους προγράμματα που λαμβάνουν το θέμα αυτό υπόψη. Πρέπει να πω ότι τα δικαιώματα, τα κοινωνικά και άλλα στις, ε, των γυναικών περιορίζονται όλο και περισσότερα. Και ενώ ε, γίνεται έκκληση στα δικαιώματα που έχουν, που τους παρέχει η θρησκεία, ό,τι γίνεται, γίνεται για να περιοριστούν τα δικαιώματα τους. Πρέπει λοιπόν να πω ότι στην Συρία, όπως και σε άλλες χώρες, η κοινωνία των ε, πολιτών υποφέρει. Θα πρέπει να είναι πολύ ε, μεγάλες οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να υποστηριχθεί η κοινωνία σύμφωνα με τις αξίες των ανθρωπίων δικαιωμάτων όπου και να είναι κανείς από τη μεριά της διεύθυνσης. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών ώστε να επωφεληθούν όλοι οι Σύριοι και όλες οι Σύριοι και να ακουστεί η φωνή του καθενός από όλους αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ε, ε, Συρίας έχει εκτός της χώρας μία άλλη προσέγγιση από αυτή που έχουμε. Υπάρχουν ε, πάρα πολύ περιορισμένα δικαιώματα για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι στη Συρία που διαρωτώνται γιατί θα πρέπει να αναλάβουν ε, να γιατί αγνοήθηκαν από την διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τόσο πολύ καιρό. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες και επίπεδο διπλωματικό. Δόθηκαν, έγιναν, δόθηκαν κάποιες ελπίδες, λήφθησαν κάποια μέτρα, αλλά οι Σύριοι πολλές φορές πιστεύουν ότι δεν ενδιαφέρει την διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση η δική τους άποψη θέλουν να έχουν η υποστήριξη. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σαφής ότι η σταθερότητα και η σταρπίση της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να γίνει και εκεί που έχει το πάνω χέρι κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την βοήθεια της, παρά το γεγονός ότι ήταν περιορισμένη, βοήθησε να γίνουν κάποια πρόοδες. Πρέπει να σας πω όμως ότι η ενεργή μεταξύ των νέων είναι της τάξης του 35% και τα θέματα τα κοινωνικά είναι για όλους πολύ δύσκολα. Κυρίως δίδεται ε, σημασία σε βοήθεια που δίδεται για την ειρηνήψη, αλλά δεν δίδεται πουθενά άλλου. Και έτσι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες για να μπορέσει να αντέξει περισσότερο ο λαός θα πρέπει να καλυφθούν από κονδύλια βοηθείας. Η πρόσβαση σε διάφορες ευκαιρίες για το λαό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό ώστε να υπάρξει ε, ανασυγκρότηση του κράτους και να περάσουμε σε μία νέα εποχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους και για να μπορέσει να υπάρξει ε, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα, προγράμματα. Βλέπουμε πόσο η ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια έχουν διασυνδεθεί σε άλλες μέρες. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν δευμέσεις εκ μέρους όλων. Δεδομένου ότι οι περισσότερες κρίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει κάνει περάσει τεχνική βοήθεια. Η στρατηγική της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να καλυφθούν οι πάντες. Αυτά στα πλαίσια των διαφόρων διαπραγματεύσεων που πρέπει να γίνουν ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση τα προγράμματα. Οι τεχνικές δεσμεύσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη το τεχνικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Η Oxfam προσπαθεί να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα και μπόρεσε να διευκολύνει πρόσβαση σε διάφορα έργα εξυγίανσης ώστε να υπάρχουν οι παροχές για όλους. Και πολλές φορές υπάρχουν τα ίδια άτομα τα οποία βρίσκουμε παντού και από τη μια μεριά και από την άλλη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι για να βοηθηθεί όλη η κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να τους κάνουμε να συμμετάσχουν σε όλες τις διασκέψεις που θα γίνουν για το μέλλον της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ένεργα για να δουν τη ζωή τους αύριο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, βελτιώσεις, πρέπει να πω ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξει περισσότερο τους Συρίους, τις γυναίκες κυρίως, τις ε, ε μειονότητες, τους ε, πρόσφυγες, τα άτομα που θέλουν να ξαναγυρίσουν στη χώρα μας. Και η κοινωνία θα πρέπει να έχει δυνατότητες πρόσβασης σε όλα τα μέσα. Χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις που υπάρχουν στην έκθεση για την βοήθεια της ε, κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι όλοι οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν εις εισόρις. Είναι θετικό αυτό το οποίο λέγεται την ισότητα των δουλειών και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σφαιρικά την κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τότση, κυρία Άνταμ. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Σας παρακαλώ να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι. Κάπου στις 3.30 περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, ο κύριος Φρόιντ είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Και θα ήθελα σε αυτό που είπε η κυρία Τότσι να σταθώ. Όταν αναφέρθηκε και ελπίζω να μην ε, αλλάξω τα λόγια σας, όταν ε, καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναδιανομή των προσφύγων. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο, ε, μία από τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναδιανομή, αλλά επίσης από το 2011 βλέπουμε την εξής αδυναμία όταν ξεκίνησαν οι σποραδικές έστω διαδηλώσεις στη Συρία. τις οποίες είχε προξενήξει λειψιδρία ή διακοπές ίδρευσης, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον από κάποια πρόσφατα άρθρα. οι Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη τη χρονική στιγμή όπου υπήρχε ακόμα δυνατότητα να αναπτύξει διάλογο και με τις δύο πλευρές, όταν ούτε Ρώσοι, ούτε Ιρανοί, ούτε Τούρκοι, ούτε Ίσης, ούτε 100.000 νεκροί, ούτε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες είχαν εμφανιστεί, αυτοί που ήρθαν δηλαδή μέχρι την Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που δεν έγινε ήταν μια συνεκτική προσέγγιση ενωμένη με αυτοπεποίθηση από πλευράς τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης αυτή που εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια πολίτες και μια σημαντική πολιτική δύναμη. Ξέρω ότι πια έσπασε το κανάτι, ε, δεν έχουμε ακόμα κοινή εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι το τελευταίο τέτοιο φαινόμενο η Συρία. Βόρεια Αφρική και χωρίς να θέλω να δώσω ονόματα, η Αλγερία είναι μία περίπτωση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διδάγματα και συμφωνείτε πως αν είχαμε μία σαφή κοινή εξωτερική πολιτική και αν υπήρχε, γιατί αυτό βλέπω να λείπει πάνω απ' όλα, ένα φορέας ο οποίο θα μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση κατά τρόπο αποτελεσματικό και να πει ότι να, στην τάδε χώρα, στη δίνα χώρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που εξελίσσεται έτσι και έτσι για να μας προειδοποιήσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν τελικά να συνέλθουμε και να αντιληφθούμε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε στην εξωτερική πολιτική για να μην μας ξεφύγει η κατάσταση τόσο όσο έχει ξεφύγει στη Συρία άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Φρόιντ. Κύριος Μπασίρ Γιούρικ Άλλος, παρακαλώ, για να κλείσω τον κατάλογο, καθώς πρέπει να προβλέψουμε και χρόνο για τις απαντήσεις των προσκεκλημένων. Μπασίρ, δύο λεπτά το πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τους ομιλητές μας σήμερα. Νομίζω ότι όλοι σήμερα ενστηριζόμαστε τη δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι η δημοκρατία συνεπάγεται και υποχρέωση λογοδοσίας. Πιστεύω ότι και οι πολίτες ε, πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους στην επιλογή, στην εκλογή της ηγεσία τους και με αυτό το ρόλο τους μπορούν και να αποφασίσουν να διώξουν από τα αξιώματα με τις εκλογές πάλι εκείνους που θεωρούν ότι δεν είναι κατάλληλοι. Κράτος δικαίου δηλαδή. Και αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου και λογοδοσία στον νόμο, η πρόοδος δεν είναι ομαλή, προκύπτουν συγκρούσεις και βέβαια οι συνέπειες της ε, απουσίας δημοκρατίας. Και το θέμα επίσης του πόσο ενστερνίζεται μια χώρα και πώς ε, ε, παίρνει στα χέρια της το μέλλον της. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε να υλοποιείται στην πράξη. Το εμπόριο επίσης έχει σημαντικό, παρά, σημαντικό ρόλο ως παράγον για την αποτυχία κάποιων κρατών της Μέσης Ανατολής. Κρατών που έχουν ε, δεχθεί εκατομμύρια προσφύγων αυτό το βάρος των προσφύγων από το Ιράκ και τη Συρία και την ε, υποσαχάρια Αφρική. Εμπόριο λοιπόν. Με το εμπόριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε το εμπόριο, τις συναλλαγές τις εμπορικές προς τις χώρες αυτές, μειώνοντας τους ε, δασμολογικούς μας, ε, τους δασμούς μας, ε, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία για τα ε, προϊόντα αυτά, δηλαδή επιτρέπονται σε παραδείγματι αντί να εξάγεται ο κόκκος του κακάο στις χώρες μας, να εξάγεται ως το τελικό προϊόν σοκολάτα από τις χώρες αυτές. Και επίσης μπορούμε να ανοίξουμε πλέον στους οριζόντες, γιατί η επιτυχία δεν χρειάζεται να προξενεί ούτε φθόνο, ούτε προσπάθεια υπονόμευσης. Μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι μιλούμε για χώρες που είναι γείτονέ μας, που μπορούμε και θέλουμε να τις βοηθήσουμε, θα χαρούμε να τις δούμε να εξασφαλίζουν την οικονομική επιτυχία. Και ολοκληρώνοντας για να κλείσω, David, θέλω να πω πως πρέπει και να υψώσουμε το παράστημα όταν κάποια κράτη υιοθετούν ανόητη στάση όπως το 2003 με τον πόλεμο στο Ιράκ, όπως με τη Λιβύη μετά. Πρέπει πιο αποφασιστικά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να πούμε ότι δεν είναι ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να προξενεί ε, ταραχές, αναταραχές και πόλεμο στη γειτονία μας. Ευχαριστώ, Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπενιφέη πολύ εύστοχα είπε ότι και εύστοχα αξιολόγησε τις ε, χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής όπου υπάρχει μερικές φορές ε, διαμάχη μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και συνήθως όταν έχουμε πρόβλημα αξιών συνήθως ε, επικαλούμαστε την ανάγκη καλής πολιτικής. Χρειάζεται λοιπόν ένας πολιτικός απολογισμός για την Αραβική Άνοιξη που μέχρι στιγμής δεν είναι θετικός. Διαπιστώσαμε πολλά λάθη και ελλείψεις στον απολογισμό αυτό. Στη Συρία έχουμε ε, πολεμική τραγωδία και μια αλληλουχία τραγικών λαθών, κατά τη γνώμη μου λόγω της αντιπολίτευσης, ε, λόγω της έλλειψης της αξιόπισης αντιπολίτευσης, αλλά έχουμε ελάθη και από την πλευρά αυτών που υποστήριξαν, ε, ε, αυτούς που υποστήριξαμε. Η Αίγυπτος, για παράδειγμα, η ε, κυβέρνηση Μούρση ε, δημιούργει πολύ περισσότερες απειλές για την ασφάλεια από ότι η κυβέρνηση Ασίσης στην Ιεμένη, που έχουμε πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή. Ένα είναι το σίγουρο, θα πρέπει να θεσπίσουμε νέα κριτήρια στην πολιτική μας. Κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πραγματική πρόοδο στην περιοχή ΜΑΒΑ και στις επιμέρους χώρες και που θα επηρεάσουν θετικά και τη δική μας ασφάλεια. Γιατί έχουμε δικαίωμα και αξίζουμε την ασφάλεια. Έχω ένα παράδειγμα, το Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν είναι χώρο που πέρασε άμεσα από τη διαδικασία της Αραβικής Άνοιξης. Πάντως η κατάσταση στο Μαρόκο σήμερα δεν είναι χειρότερη από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ποιος σε αυτή την περιοχή είναι φίλος χώρα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τους φίλους μας και να στηρίζουμε τους φίλους μας, τις φιλικές χώρες. Επίσης θα πρέπει να δείξουμε και μια φαντασία και να δούμε τι αρνητικές αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν κρίσεις και θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν και από τα παθήματά μας για να αποφύγουμε στο μέλλον ε, επανάληψη της δραματικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα στη Συρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά για να απαντήσετε. Παρακαλώ, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Να το αντιστρέψουμε τη σειρά. Ωραία. Ladies first, κυρία Τότσι. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομη για να δώσω απαντήσει σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν. Συμφωνώ απολύτως με την ε, εκτίμηση πω χρειάζεται ενότητα. Βεβαίω, ε, και αποτελεί αφετηρία για οτιδήποτε πράκτουμε. Είτε σε αυτή την περιοχή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη. Αλλά για να ε, κοιτάξουμε πίσω και σε σχέση με τη Συρία, και το παράδειγμα που επισημάνθηκε, το λάθος μας τότε ήταν, άλλωστε είναι και πολύ συχνά το λάθος μας αυτό, ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση τίνουμε να κλειδονιζόμαστε, να ραντεβόμαστε κατά τρόπο αρκετά ακραίο θα έλεγα και δραματικό ανάμεσα σε, στα άκρα της ύβρεως αφενός ή της υπερβολικής ταπεινοφροσύνης αφετέρου. Το 11 λοιπόν το λάθος που μας οδήγησε στο να μην κάνουμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, δηλαδή να αρχίσουμε τις συνομιλίες αμέσως με τον καθέναν, ήταν ότι θεωρούσαμε πως μπορούσαμε να κερδίσουμε. Εμείς η Δύση. Ε, θεωρώντας ότι να είχε ήδη καταρρεύσει το καθεστώς του Μπεναλή, ο Μπουμπάρα ε, και, άρα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε με κανέναν, να μην συνομιλήσουμε κανέναν, αλλά απλώ πιέζοντας ε, από τη δική μας πλευρά βέβαια να κερδίσουν αυτοί που υποστηρίζαμε, χωρίς όμως να κάνουμε και ό,τι χρειαζόταν για να επικρατήσουν αυτοί θα μπορούσαν αλλά και πάλι το, τα γεγονότα μετράνε και Ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η αδυναμία ότι επαναπαυόμενοι, χωρίς να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια από τα ζητήματα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως επισημάνθηκαν και νωρίτερα, να θέσουμε τα ζητήματα, δηλαδή ανοικοδόμηση μετά από μια σύγκρουση που πολιτικά προξενήσαμε, έτσι, όχι στρατιωτικά γιατί δεν κάναμε βομβαρδισμούς, αλλά που χάσαμε πολιτικά. Πρώτη φορά μας απασχολεί ένα τέτοιο ερώτημα, χωρίς να ρωτάμε, να μην θέτουμε αυτά τα, χωρίς να θέτουμε αυτά τα σκληρά ε, ε, ερωτηματικά. Άμα δεν τα θέσουμε όμως αυτά με ερωτηματικά, δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε μια σύγκρουση στρατιωτική, στην οποία έχουμε επιλέξει να, να υποστηρίζουμε τη μία πλευρά. Άρα και συμφωνώντας ε, απολύτως με την εκτίμηση πως χρειάζεται ενότητα, εγώ θεωρώ ότι αφενός η αδυναμία, αφετέρου η, η δηλαδή αυτή η σχιζοφρενή στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αιτία των αποτυχιών μας. Ευχαριστώ πολύ για να δώσω και εγώ απάντηση στο ζήτημα της ε, συνοχής ή ενός κοινού οράματος που δεν έχει η ευρωπαϊκή πολιτική η Συριακή, για να μιλήσω και για στρατιωτική προοπτική. Ανοικοδόμηση. Πολιτικό βέβαια ζήτημα. Ως ανθρωπιστικός ε, φορέας εμείς δεν ασχολούμαστε με την ανοικοδόμηση. Αλλά καθώς η ανοικοδόμηση είναι πολιτικό ζήτημα. Και καθώς υπάρχουν και τόσοι περιορισμοί στην ανάπτυξη των μέτρων και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διστακτική στην ανάπτυξη του θέματος και τη συζήτηση του θέματος της ανοικοδόμησης για την ανθρωπιστική πτυχή αυτό έχει σαν συνέπεια πώς περιορίζεται το πεδίο για ανθρωπιστική παρέμβαση. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την κατάσταση στη Συρία με άλλες πάλι ανθρωπιστικής κρίσης, βλέπουμε ότι αμφισβήτηση ως προς την ανθρωπιστική πρόσβαση δεν υπάρχει. Δηλαδή, και η διάσωση ζώων και η ε, ανάκτηση, η διάσωση από περιοχές επικίνδυνες υπάρχουν στις υπόλοιπες ανθρωπιστικές κρίσεις, ενώ στη Συρία η ίδια η ανθρωπιστική παρέμβαση δεν μπόρεσε να πάει περαιτέρω της διάσωσης ζωών. Και καθώς συνεχίζεται εδώ και 8 χρόνια αυτό, αυτή η σύγκρουση, δεν μπορεί να είναι σε αυτού του τύπου η βοήθεια όσο θα όφιλε να είναι. Στην έγκαιρη διάσωση των ανθρώπων αυτών ή την ε, δυνατότητα εκένωσης των περιοχών τους. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ή περιοχές που εξαρτώνται 100% από την ανθρωπιστική βοήθεια. Πάλι δεν γίνεται τίποτα. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει αυτούς τους πληθυσμού. Ε, πληθυσμούς. Και, και στην ανοικοδόμηση, δηλαδή στην ανάκτηση των δυνατοτήτων διαβίωσης, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται απόλυτος από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τότσι, κύριε Μουτάζ Αντβάμ και για το τελικό λόγο να ολοκληρώσουμε. Φυσικά θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπενιφέη. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να πω πως σύντομη ένα αλλά και πολύ εντατική ανταλλαγή απόψεων η σημερινή και μας δίνει πολύ υλικό για να συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Τονίζω τα λόγια της κυρίας Τότσι και την αναφορά στο, στα συμβουλευτικά συμβούλια που αναφέρουμε και στην έκθεση. Προτείνω λοιπόν και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας, να μην περιοριστεί η δυνατότητα για ανάπτυξη του, των δραστηριοτήτων τους Επίσης η προσέγγιση μας, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κύριος Αντάμ επίσης. Μας είπε ξεκάθαρα πιστεύω, καθώς γνωρίζει επιτόπου την ε, κατάσταση και την ανάγκη για περισσότερη ανάπτυξη ε, δυνατοτήτων ε, κοινωνίας των πολιτών, δικαιωμάτων των γυναικών και γενικότερα δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των γυναικών που ιδιαίτερα τονίσαμε εμείς και στην έκθεση έχοντας εξετάσει διάφορες χώρες και τα καθεστώτα τους, αλλά ιδιαίτερα τη Συρία, αλλά και την περαιτέρω συνέχεια που θα δοθεί, ε, το, να μην επιβάλλονται δηλαδή μόνο κυρώσεις ε, σαν κάτι το μεμονωμένο, αλλά να υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση και συνέπεια, συνοχή στη δράση μας. Αυτά λοιπόν όλα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, τον πρόεδρο, τους συζητητές, την κυρία Τότσι και τον κύριο Άνταμ για την ευκαιρία για την ανταλλαγή αυτή απόψε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε. Καλή τύχη και καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε και να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, με το σημείο 31 δηλαδή, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα. Ησυχία παρακαλώ ήθελα να τραβήξω και την προσοχή των σοσιαλιστών και δημοκρατών προ τον σοσιαλδημοκράτη καλεσμένο μα. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ρουμανία, τον κύριο Τέοντορ Μελεσκάνου. Όπω ξέρουμε, η πατρίδα του έχει αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου. Έχουμε πολλού συναδέλφου από τη Ρουμανία που παρίστανται εδώ. Φυσικό είναι και αναμενόμενο. Θα Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά λοιπόν και στα ρουμανικά ο πρόεδρος. Συνάντησα τον Υπουργό Μελεσκάνου στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα και μιλά από αρκετές, αρκετές γλώσσες. Μιλάει άψογα αγγλικά, γαλλικά, φυσικά και ρουμανικά. Τον συνοδεύουν η κυρία Ριμενίτα Οντουβέσκου, μόνιμη αντιπρόσωπος της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ήρθατε και ο κύριος Στέφαν Τίντσα, Τίνκα, πολιτικός διευθυντής. Καλώς ήρθατε. Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα μέλη της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες, το κάναμε και στο Στρασβούργο Μας ενδιαφέρει η πολιτική διεύρυνση, προστατικά Βαλκάνια, Τουρκία, διατλαντικές σχέσεις, κατάσταση στη Ιράν, Βόρεια Κορέα, κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Επίσης θα έχει δύσκολη προεδρία Ρουμανία πρώτον λόγω των ευρωεκλογών και δεύτερον θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις βεβαιότητες που εγείρει το Brexit σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελικά το Brexit. Δύσκολη και απαιτητική προεδρία λοιπόν. Πάντω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρεί στα θέματα που αφορούν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το, το Μηχανισμό Γειτονία Ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία και το νέο προταξιακό μηχανισμό IPA3. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση και για τα δύο θέματα πριν το τέλο τη κοινοβουλευτική ε, σας καλωσορίζουμε. Θα σας βλέπουμε συχνά τους υπόλοιπους 5,5 μήνες της Ρουμανικής Προεδρίας και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση εκπροσωπώ το μικρότερο τμήμα του κυβερνητικού συσχηματισμού. μέλος της Συμμαχίας ε, Φιλελευθέρων και Δημοκρατών και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας παρουσιάσω τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, νιώθω μεγάλη χαρά και νιώθω την προνόμιό μου που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας, που εσαρκώνει την θεσμική εταιρική σχέση στην οποία από κοινού Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν του στόχου εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκα πολύ από την επιτροπή σα. Και όταν προσπάθησα να την παραλύσω με την Επιτροπή Εξωτερικών τη Ρουμανική Βουλή, διαπίστωσα ότι ε, έχουμε μεγάλη διαφορά ε, στον αριθμό των μελών. Αλλά αυτή είναι η διαφορά Ρουμανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, θα μιλήσω σήμερα εκ μέρους μιας χώρας που βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έβλεπε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, σύμβολο της ε, υλοποίησης της υπόσχεσης δημοκρατίας, ευημερίας και ασφάλειας. Καθοριζόμαστε από τις επιλογές μας. Επιλέξαμε λοιπόν να, μείνουμε, να είμαστε ενωμένοι υπό την ίδια σημαία και αξίες, τους κοινούς στόχους και αξίες που έχουμε με τους στενότερους φίλους μας. Και ως κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρουμανία ανέκαθεν ε, ε, συνειδητοποιούσε την ανάγκη να αναλάβει τις ευθύνες της και να εξυπηρετήσει το στόχο της καλύτερης Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που μας δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία μας να αναλάβουμε την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Και κατά την έναρξη της Προεδρίας διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Έχουμε τον Brexit, τις ευρωεκλογέ τις ε, διαπραγματεύσεις για βασικές πολιτικές και στρατηγικές ε, εμβληματικού χαρακτήρα, όπως είναι το στρατηγικό σχέδιο δράσης για μετά το 2019, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυστυχώς το διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα η πραγματικότητα που περιστοιχίζει την Ευρώπη ε, περιέχουν πολλές προκλήσεις. Όλες αυτές οι προκλήσεις ενώ βρισκόμαστε στο επίκεντρο της ε, θεμελιώδους συζήτησης ε, της μελλοντικής μας πορείας, ε, μας βρίσκει σε μια εποχή που καλούμαστε να κάνουμε σημαντικές επιλογές. Και οι στόχοι της Προεδρίας μας αντανακλούν όχι μόνο τις φιλοδοξίες μας για τη θητεία μας αυτή και για την εντολή μας αυτή, αλλά και για, την, για το όραμά μας για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση και από και από εξωτερικής κοπιάς. Και από αυτή την προοπτική η Ρουμανική Προεδρία θα θέσει τη συνοχή στο επίκεντρο του προγραμματός της. Και θεωρούμε ότι η συνοχή είναι η έκφραση της ε, επικοδομητικής όθησης ε, των χωρών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς μια οικονομική, κοινωνική και πολιτική πρόοδο. Γι' αυτό και το σύνθημα της Προεδρίας είναι συνοχή η ευρωπαϊκή κοινή αξία. Το θεματολόγιο μας για τους επόμενους μήνες ε, θα επικεντρώνεται σε τέσσερις διαστάσεις. Σε περισσότερη σύγκληση, σε ασφαλέστερη Ευρώπη, σε ισχυρότερη θέση παγκοσμίω και σε πιο στιβαρές και κοινέ αξίες. Ε, είναι αυτονόητο ότι η εξάμεινη εντολή μας είναι μόνο μία πινακίδα στο μακρύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Ε, τα θεμέλια και η εγγύηση οποιασδήποτε επιτυχίας είναι η, η συνέχεια και το απάφγασμα μακροπρόθεσμων και μακροχρόνια προσπαθειών. Εξού και η σημασία της ε, θεσμικής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσαρκώνει την ίδια την ιδέα της ευρωπαϊκής νομοποίησης. Και ελπίζω να έχουμε στενό διάλογο γιατί έχουμε κοινό, ε, κοινή κατεύθυνση και κοινό μέλημα τους πολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώνουμε τις προσπάθειές μας και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή σας, την ΑΦΕΤ και με τους ε, ευρωβουλευτές ξεχωριστά, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τους περιορισμούς ε, λόγω των επικείμενων εκλογών του Μαΐου. Βεβαίως ακριβώς σε αυτή την ε, προεκλογική στιγμή θα πρέπει εμείς οι πολιτικοί να ενημερώσουμε τους ψηφοφόρους μας, εκλογικές μας περιφέρειες για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας και στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ό,τι αφορά τις προτεραιότητες για την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής δράσης, θα ήθελα να σας αποκαλύψω και τις δεξιότητες μου στα γαλλικά, μιλώντας γαλλικά, όντως φόρος τιμής προς τη γλώσσα αυτή και εκφράζοντας την πολύτιμη πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το τρίο των Προεδριών, τη Φιλανδία και την Κροατία, συμφωνήσαμε στο πρόγραμμα του τρίο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω πρόοδο κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής. Μεταξύ άλλων, κοινέ μας προτεραιότητες ε, συμπεριλαμβάνουν ε, η δέσμευσή μας προς τη διεύρυνση, η πρόθεση πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ της Ένωσης και των γειτονικών της χωρών, προς Ανατολάς και προς τον Νότο, ενίσχυση και διαφύλαξη του πολυμερού συστήματος βάση κανόνων στα πλαίσια του ΟΗΕ, με ενίσχυση των συνεργατικών ε, περιφερειακών τάξεων και της διατλαντικής σχέσεις, προωθώντας ε, το έργο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας με αποτελεσματικές ε, και εύρυθμες μεθόδους. Μια και είμαστε η πρώτη Προεδρία από τις τρεις, το Εθνικό Πρόγραμμα Εργασιών βάζει τα θεμέλια για τη συγκεκριμενοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. Με τόλμη και ενθουσιασμό, κατά την πρώτη Προεδρία μας, Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά την ύπατη εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές και συνεκτικές εξωτερικές δράσεις. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια καρποφόρο συνεργασία με την ΕΕ και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, ε, το παγκόσμιο προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα εξαρτηθεί ιδιαίτερος από το ρυθμό με τον οποίο εφαρμόζουμε την παγκόσμια στρατηγική μας και από την αποτελεσματικότητα των επιμέρους μηχανισμών της. Πρόσφατα αναπτύξαμε εργαλεία για την διαμόρφωση και την πρόθεση του ευρωπαϊκού τρόπου κατά την αναζήτηση ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Η αποτελεσματικότητα, μία από τις τέσσερις προτεραιότητές μας, θα πρέπει να αφορά και τους πόρους, αλλά και το τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η αποτελεσματικότητα θα είναι το ζητούμενο και στην κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ενισχύοντας και τη σκληρή και την ήπια δύναμη της Ευρώπης. Υπάρχοντας μηχανισμοί, όπως συντονισμένη της αξιολόγηση της Εθνικής Άμυνας, ο μόνιμος διαρθρωμένος, ε, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα πρέπει να ενισχυθούν και εξασφαλίζοντα τη συνοχή τους ταυτόχρονα με παρόμοια εργαλεία του ΝΑΤΟ και παρόμοιε διαδικασίε στο ΝΑΤΟ. Θα στηρίξουμε και τις ερευνητικές δράσεις και δράσεις τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και του βιομηχανικού τομέα άμυνας. Τέτοιου είδου πρόοδο δεν θα πρέπει να γίνει ει βάρο του πολιτικού σκέλου τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Αντίθετα, η πρόθεση συνεργασίας μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου είναι απαραίτητη και μάλιστα θα προωθήσουμε την εφαρμογή του νέου σχεδίου πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σφαιρική προσέγγιση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου συγκρούσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια σφαιρική και ελαστική απάντηση και στο πολιτικό σκέλος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Επίσης θέλουμε ρωμαλές, στιβαρές ε, διατελετικές σχέσεις. Η διατελετική εταιρική σχέση είναι σημαντικότερη από ποτέ. Η αξία και το παρελθόν των σχέσεων μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά δείχνουν προς παρόμοιες σχέσεις και στο μέλλον. Θα πρέπει να βρούμε έμπνευση και για να συνεχίσουμε να γεφυρώνουμε τα μεταξύ μας κενά. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα, να καταπολεμήσουμε τις υβριδικές απειλές και να διευρύνουμε τις ικανότητες στρατηγικής επικοινωνίας μας βάσει μια σφαιρική προσέγγισης που θα καλύπτει και τους τρεις τομείς. Θα διδαχθούμε από τα μαθήματα της συνεργασίας με τους εξωτερικούς εταίρους και θα αντιλήσουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα για την ασφάλειά μας και από εσωτερική και από εξωτερική άποψη. Θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση στις πιο ευάλωτες στιγμές και θα ενισχύσουμε την αθεκτικότητα της κοινωνίας από πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα προς πιο μακροπρόθεσμες πολιτικές. Επίσης, κατά την αναζήτηση αυτής της αποτελεσματικότητας, συζητώντα το επίπεδο φιλοδοξίας της ευρωπαϊκής δράσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις διαφορετικές επιλογές ή βλέψεις ε, και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της συζήτησης για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ρουμανική Προεδρία θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής διαδικασίας για την εξωτερική συνιστόσα του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και για τη μελλοντική χρηματοδότηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα. Και αυτό θα είναι η λιδία λίθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πια χωρών. Έχουμε επίγνωση ότι η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερη προτεραιότητά μας αφορά τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ορόσημο της διαδικασίας διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπό αυτό το πνεύμα, τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε ε, μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Ελπίζουμε ότι η κοινή μας ε, υποστήριξη μαζί με την ε, ανάληψη ευθύνη και από του εταίρου μα ε, για συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα που είναι απαραίτητε προποθέσει για οποιαδήποτε διεύρυνση, θα δημιουργήσουν ένα πολύ πρόσφορο έδαφο ώστε να αποφασίσει και το Συμβούλιο να ξεκινήσει ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη ΦΥΡΟΜ και την Αλβανία τον Ιούνιο του 2019. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη επίση θα πρέπει να ε, λάβουν την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντα μία ε, άνηση προσέγγιση και χωρί ισορροπία στην περιοχή. Πέραν της ε, διαδικασίας διαβρύσης, η περιφερειακή πραγματικότητα απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό μυαλή προσέγγιση και ευρύτερη συνεργασία και από αυτή την άποψη θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία των Δυτικών Βαλκανίων δίνοντας ενάβησματα για μια δραστήρια ενεργή ηθαγένεια και μια παιδεία αμοιβαία κατανόησης και διαλόγου. Επίσης θα, θα ρίνουμε ε, συζήτηση για το πώς θα δώσουμε προτεραιότητα στην περιφερειακή συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και κυρίως για το κατά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμμετέχει σε διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες και δομές. Έρχομαι τώρα στην Τουρκία. Συνολικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε ανοιχτή αυτές της διάβλους επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη, τους διάβλους επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια υποψήφια χώρα και στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς. Και φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιληφθεί τη ιδιαίτερη προσοχή που δίνει η Ρουμανία στην Τουρκία, γιατί και η Ρουμανία είναι χώρα του περιοχή της περιοχής του Ευξηνοπόντου και έχουμε επίγνωση της στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, η Ρωμανία ε, θα θέσει την ανατολική γειτονία ε, ως εμβληματικό κλάδο και προτεραιότητα της Προεδρίας της. Το Μάιο του 2019 θα εορτάσουμε την δέκατη επέτειο των, της θέσπισης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης του 2009 και αυτήν την άποψη θα επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας ώστε αυτή η επέτειος να χαρακτηριστεί από αισθητή πρόοδο στην εξέλιξη των σχέσεων με τους εταίρους μας και στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων για το 2020. Ταυτόχρονα θα διοργανώσουμε μια συζήτηση για το μέλλον της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης μετά το 2020. Και αυτή η δεκαετής πολιτική ήδη ε, έχει δώσει μέλλον, μελλοντική προοπτική στους ανατολικούς εταίρους μας και θα είναι σημαντικό όχι μόνο να εκλεπτήσουμε την ανατολική εταιρική σχέση, αλλά ταυτόχρονα οι χώρες αυτές να συνεχίσουν το δρόμο τους προς την Ευρώπη. Και από αυτή την άποψη οι δύο ε, ε, επικείμενες εκλογές στη Μολδαβία και στην Ουκρανία θα λάβουν ιδιαίτερη σημασία, στρατηγική θα έλεγα, και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ε, στρατηγική σημασία για τη Ρουμανία θα έχει η επαναφορά της Μαύρης Θάλασσας στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Και αυτή θα είναι η σημαντική μας προτεραιότητα. Ε, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα σχέδια και τομέακή συνεργασίας ε, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας γύρω από τον εύξηνο πόντο, στην έρευνα και την καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. Ε, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγύψουμε περισσότερο σε πολυδιάστατα τομεακά ζητήματα και σε ένα πικοδομητικό θεματολόγιο που θα, δώσει, θα αναζωογονήσει τη συνέργεια της Μαύρης Θάλασσας και θα ε, δώσει τον μελλοντικό προγραμματισμό θα δώσει στο μελλοντικό προγραμματισμό ένα πιο βιώσιμο χαρακτήρα. Μια άλλη περιοχή προτεραιότητα για μα θα είναι η περιοχή τη κεντρική αξία, που είναι σημαντικό σημείο ζεύξη μεταξύ τη Ευρώπη και τη Ασία. Και μάλιστα ε, μετά την πρόσφατη έγκριση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνδεσιμότητα με την Ασία και αναμένοντας τη μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, η Προεδρία μας θα συμβάλλει στο να ε, αναζωογονηθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής αυτής της Κεντρικής Ασίας. Και θα επεκτείνουμε τη σφαίρα των ενδιαφερόντων μας ε, στην πολυμέρεια και στην, παγκόσμια τάξη βάση κανόνων. Και παρά τις ε, παλιές και νέες βεβαιότητες, αυτή η δέσμευση υπέρ της ε, πολυμέρειας βάση κανόνων θα είναι δική μας πεποίθηση και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε θετικές δυνάμεις αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο και η εφαρμογή της, θεματολογίου τη αηφόρου βιώσιμη ανάπτυξη και η συνεργασία στα θέματα διατήρηση ειρήνη και αθεκτικότητα σε καταστροφέ θα είναι βασικά θέματα τη Προεδρία. Όπω είπα και στην αρχή τη παρέμβασή μου, το πρόγραμμα εργασιών τη Ρουμανική Προεδρία περιστρέφεται γύρω από τέσσερι άξονε. Την Ευρώπη της σύγκληση, την Ευρώπη της ασφάλειας, την Ευρώπη ω παγκόσμιο παράγοντα και την Ευρώπη των κοινών αξιών. Βέβαια, η έκτακτη διάσκεψη κορυφή του Συμπίου, δεδομένου του ρόλου της για, το για, το... για τη διαμόρφωση της μελλοντική στρατηγικής, μας υπενθυμίζει και έναν πέμπτο άξονα, την Ευρώπη που ε, θέλει και οφείλει να επιλέγει μόνη της και για τον εαυτό της. Και η Ρουμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψε. Thank you, Minister presenting the... Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Προς το παρέλ έχουν ζητήσει το λόγο 11 συνάδελφοι. Πολύ καλή αρχή λοιπόν. Έχουμε 35 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρακαλώ λοιπόν ο κάθε συνάδελφος να λάβει το λόγο για δύο λεπτά ώστε να έχει αρκετό χρόνο ο υπουργό για να απαντήσει. Ε, εσείς, εσείς σφαιρικά κύριε Υπουργέ μπορείτε να έχετε 10 λεπτά η απάντηση. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον κύριο Πρέντα, στον συνάδελφο από τη Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην ε, Προεδρία. Υπάρχουν τρία στοιχεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Πρώτα απ' όλα, οι πρόσφατες ε, παρατηρήσεις του Κινέζου Πρόεδρου Τσίζι Πινγκ για την δυνατότητα επανένωσης της ε, Κίνας με την ένταξη στην Κίνα πλέον της Ταϊβάν. Ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι θα πρέπει κάτι να, θα πρέπει κάτι να πει και το Συμβούλιο για τέτοιου είδου θέματα. Δεύτερον, η κυβέρνησή σας πολλές φορές ανέφερε ότι θα σκέφτεται τη μετεγκατάσταση της ε, πρεσβείας σας στην Ιερουσαλήμ λάβετε υπόψη την γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Τρίτο θέμα, Μολδαβία. Πριν από την Προεδρία, το Βουκουρέστι μπλόκαρε κάποια συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου ε, που αφορούσαν τη Μολδαβία. σε σχέση με την κατάσταση της δημοκρατίας στη Μολδαβία και κάποιες παρατηρήσεις που έκανε η είπατε εκπρόσωπος. Και βεβαίως ο κύριος Πλάχινουκ δεν ήταν ευτυχής με τις εξελίξεις και με αυτά τα οποία είπε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι, κάποιες αποστολές ε, μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου στη Μολδαβία. Σκέφτεστε να οργανώσετε εξ ονόμου της Ευρωπαϊκής για να δείτε τόπου τι γίνεται. Ευχαριστώ, Χριστιαν. Πρόεδρος Κριστέα. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Υπουργό. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Πρώτα απ' όλα, η Ρωμανία έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τη σχέση με τη Μολδαβία πραγματικά τι περιμένετε μετά από τις εκλογές, τις βουλευτικές που προβλέπουν το Φεβρουάριο στη Μολδαβία. Υπήρξε μια συνάντηση υπουργική ε, χθες το πρωί Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίσαμε εμείς για συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Τον επόμενο μήνα θα γίνουν πάρα πολύ σημαντικές διαπραγματεύσει για θέματα ελεύθερου εμπορίου με τη Σιγκαπούρη. Ποια είναι η θέση σας ως υπουργό όσον αφορά την ε, βελτίωση αυτών των σχέσεων και την αναβάθμισή τους με έναν σημαντικό εταίρο τόσο σημαντικό. Και τώρα, φτάνουμε στον Τζολ Τάνοκ που είναι φίλος των Ρουμάνων. Ναι, ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στον Υπουργό Διαδικαστικό. Καταρχάς, η Προεδρία έχει να κάνει βέβαια με τη διεύρυνση και με την πολιτική της γειτονίας μπορεί υπό την ιδιότητά σας ως Υπουργό των Εξωτερικών να σας ενδιαφέρει και το θέμα της Ταϊβάν, της Κίνας κτλ. Αλλά ω εκ τη συνθήκης ρόλο σα είναι μόνο αυτή η τομή τη εξωτερική πολιτική. Τα λοιπά είναι τη αρμοδιότητά, τη είπα τη εκπροσώπου, οπότε αντιλαμβάνομαι εγώ. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερος για την προσήλωση στην ε, πολυμερή συνεργασία και βέβαια την καταπολέμηση των εθνικισμών στην Ήπειρό μας και Αλαχού για τη Ρουμανία που παραδοσιακά θα θεωρούνταν βαλκανική χώρα. Είμαι μάλιστα εισηγητής ε, τουλάχιστον για το προσεχές εξάμεινο για το Μαυροβούνιο και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλιά σας που υποστηρίζουν την προσχώρηση του Μαυροβουνίου και της ε, Σερβίας για την ε, Μακεδονία που πρόκειται, λέει ο να γίνει δημοψήφισμα και Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα ε, και να προχωρήσει. Αυτό θα έχει βέβαια συνέπειε και για την ε, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Η Ουκρανία, η συμφωνία των Μπάσκ και Μίνσκ ε, είναι πολύ σημαντικές και ελπίζουμε να, να δοθεί συνέχεια. Όλα αυτά είναι θέματα μεγάλης σημασίας και για την πατρίδα μου και ενώ του Brexit. Ίσως εσείς χρειαστεί την ε, ημερομηνία της ε, εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου να την διαχειριστείτε εσείς. Εκτός και αν δοθεί παράταση στο Brexit, πράγμα για το οποίο δεν θα σας καλέσω να σχολιάσετε γιατί ίσως να μην θέλετε. Αλλά μπορεί και αυτό να συμβεί. Κυκλοφορεί στις ειδήσεις, σε πάση περιπτώσει. Πάντως μια έκκληση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη κυβέρνηση του να παραμείνει στην πρίζα ούτως πιν για να μην αποκοπεί από τις εξελίξεις κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και ταυτόχρονα σε συνεργασία με την ΠΕΣΚΟ και την CSTP, την ΚΕΠΑ δηλαδή, την ειδική ε, σχέση και συνεργασία για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Μεγάλη πρόκληση, ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν υπάρξει καμία συμφωνία για τον Brexit και άρα δεν υπάρξει και μεταβατική περίοδος για τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Ρεμπέκα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ μου άρεσε η υπόσχεση ότι θα εστιαστείτε στην Επιτροπή, στην στρατηγική γειτονία και της... Ε, οι γειτονικέ και συνδεδεμένε χώρες. Έχω μια ξεκάθαρη ερώτηση, ειλικρινή ερώτηση. Όλες αυτές οι χώρες συνδεδεμένε και τα λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα που είναι η διαφθορά. Η Ουκρανία, παραδείγματι, όπου μαζί με τους Ουκρανούς ε, χτίσαμε την εισαγγελία για την πάταξη τη διαφθορά. Ακολουθώντας και το παράδειγμα της Ρουμανίας ε, για την ε, ειδική εισαγγελία αυτή κατά της διαφθοράς, αλλά βέβαια εδώ πρέπει να συζητήσουμε και το ζήτημα ακουβιζή στην Ρουμανία και των όσων ακολούθησαν. Ε, ρωτώ λοιπόν ως υπόδειγμα στη γειτονία, τι ρόλο μπορεί να δραματίσετε εσείς ως ε, Ρουμανία, ως υπουργό Εξωτερικών, θέλω να μου το πείτε, για δε την Τουρκία. Θα συζητήσουμε βέβαια στην προσεχή περίοδο την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η εισηγήτρια στο σχέδιο εκθέσεως καλεί να αποφασιστεί η άρση των συνομιλιών. Θεωρείται ότι ο κίνδυνος για εμφύλιο πόλεμο στην Τουρκία ο κίνδυνος για παρέμβαση στρατιωτική της ε, Τουρκίας στη Συρία σημαίνει για τη χώρα αυτή που όχι μόνο είναι υποψήφια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέλος του ΝΑΤΟ μπορούν να συνάδουν με την προοπτική για ένταξη. Ευχαριστώ πολύ Ρεμπέκα Χάρμς. Κύριε Σκουκάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στο επόμενο εξάμεινο για σας, για την αναφερθήκατε λοιπόν στις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και βέβαια εδώ και καιρό εδώ μιλάμε με πολύ ενθουσιασμό για τη διεύρυνση, στρατηγική της διεύρυνσης με την Βουλγαρική Προεδρία που ήταν πολύ φιλόδοξη να πιέσει για περισσότερη διεύρυνση, πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής μετά από 15 χρόνια, Αυστριακή Προεδρία με τόσες γνώσεις και εξειδίκευση στα θέματα της διεύρυνσης που ε, είχε και εν τέλει ο απολογισμός ήταν ισχνός. Λυπούμε λοιπόν, που σας το λέω έτσι λοιπόν. Γιατί όλοι λέμε «Αχ, χρυσή ευκαιρία για τα Δυτικά Βαλκάνια». Βουλγαρία αφενό, Αυστρία αφετέρου και έρχεται και η δική σα η Προεδρία. Ε, ξέρουμε ότι ήσασταν κάπως πιο επιφυλακτικοί. Εξαιρετική ευκαιρία λοιπόν σα δίνετε να του ξαφνιάστε όλους όσοι ήταν επιφυλακτικοί απέναντί σα. Να του κάνετε να μιλούν για εσά όλο ο κόσμο γιατί φοβούμαι ότι χάνουμε την αξιοπιστία μας στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί εμείς τους λέμε τι προϋποθέσεις έχουν να πληρώσουν, τις πληρούν, αλλά μετά διαφωνούμε. Και ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι χώρες. Αλλά δεν μπορώ να το πω και ανοιχτά. Ξέρετε λοιπόν ότι όλοι θα κοιτούν με το φακό, με το μικροσκόπιο να δούνε πώς θα τα καταφέρετε. Παρακαλώ, ξαφνιάστε τους λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Πάσκου. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. στην πολιτική απαραίτητα είναι τα πάντα, τα πάντα όμως είναι και ανεπαρκή. Αυτό κύριε Κούκαν για σας. Ας αλλάξω όμως εγώ λίγο κατεύθυνση και ας ρωτήσω τον Υπουργό. Τι φρονεί για την πολιτική σημασία της συμπερίληψης της χώρας του το νομίσματός του στην Ευρωομάδα ενισχύει περισσότερο τη χώρα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Τούκες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπουργέ, Έχει τώρα την Προεδρία η Ρουμανία, έχει ορίσει τους στόχους της. Ευρώπη καλύτερη, Ευρώπη πιο ενωμένη. Συνοχή λοιπόν σε συγκεκριμένους όρους. Μείωση των ε, διαφορών μεταξύ των κρατών κτλ. Στόχοι ευρωπαϊκοί λοιπόν, στόχοι που και εμείς δεν έχουμε ακόμα επιτύχει. Και οι πολιτικοί βλέπουμε ότι δεν ήταν διχασμένοι ποτέ όσο τώρα. Βλέπουμε να αναδεικνύεται και ένας ε, ουγγρικός εθνικισμός στη Ρουμανία. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορεί η χώρα μας να βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα και να εξασφαλίσουμε τους στόχους της συνοχής, της συνένεσης, της ομόνιας. Όταν η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Για να μην εξάγουμε τα προβλήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι. Και κάτι ακόμη. Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας τον κρατών που προχώρησε με, πολλούς, ε, με πολλές συναντήσεις και με τον ομολογό σας της Ουγγαρίας με δηλώσεις και διακηρύξεις όπου λεγόταν ότι επικρατεί αμοιβαίος σεβασμός και στο στόχος είναι η ισότιμη συνεργασία. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ ωραία. Ωστόσο βλέπω ότι οι, οι, οι ευρωβουλευτές της δικής σας πολιτικής οικογένειας που ανήκουν στο Άλντε, οι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές, καταψήφισαν την έκθεση Αργεντίνη που θα ενθάρρυνε μια τέτοια συνεργασία. Πώς τη βλέπετε λοιπόν εσείς αυτή την ουγγρο-ρουμανική συνεργασία, κυρίως για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ευχαριστώ κύριος Φροντζούλικα. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Αναφέρατε πολλές φορές ότι η Ρουμανία θεωρείται είναι πολύ σημαντική η πολιτική διεύρυνση. Αλλά βεβαίως αναλαμβάνει και πολύ ισχυρίζοντας μέσα όσον αφορά την ε, ε, ανατολική εταιρική σχέση. Πώς λοιπόν υποστηρίζεται τις προσπάθειες που καταβάλουν οι εταίροι μας ε, στην Ανατολή. Κυρίως και τις χώρες οι οποίες έχουν συμφωνίες, χώρες όπως Μολδαβία ή άλλες. Κύριε Υπουργέ, το Συμβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητα μεταξύ των κρατών. Πώς μπορούμε εμείς να στείλουμε και μήνυμα που υπάρχει εκ μέρους κάποιων πολιτικών ότι υπάρχουν πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας πολίτες. Πώς μπορείτε να κάνετε εσείς κάτι κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν Μόν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν με πλήσει η σημασία που θέλετε να αποδώσετε στα θέματα της γειτονία. Μιλήσατε μόνο για την ε, ανατολική γειτονία. Είναι σημαντικό αυτό βέβαια για τη Ρουμανία, αλλά πιστεύω ότι η μεσογειακή γειτονία στο Νότο επίσης είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι Ισπανός και πολλές χώρες ευρωπαϊκές είμαστε γείτενες των λαών που ζουν νοτίως τη Μεσογείου. Θα ήθελα λοιπόν και για αυτή την ε, διάσταση της γειτονία να μιλήσει τη Μεσογειακή. Και δεδομένου ότι έχω το λόγο θα ήθελα να σας πω το εξής. Μιλήστε για τη Βενεζουέλα, που ζει δραματικέ στιγμέ. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί το προσέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα. Το, το Συμβούλιο όμω θα πρέπει το ίδιο Και επίση, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν και διαπραγματεύσουν το Μερκοσούρ. Διότι είναι σημαντικό αυτό για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι εμπορικές μας σχέσεις. Μακάρι λοιπόν να μπορέσετε να δώσετε μια νέα όθηση στο θέμα αυτών των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες, σας καλωσορίζω. Κύριε Υπουργέ, η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος είναι κάτι το οποίο αφορά επίσης την τρομοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για σας. Είναι κάτι το οποίο το αφήνετε στα χέρια των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που είναι δικό τους θέμα, θέμα αποκλειστικά ή σας αφορά και εσάς, γιατί έχει και πολιτική διάσταση. Επίσης, η... μας είπε η νεοεκλεγής πρόεδρος της Γεωργίας ποιες είναι οι προσδοκίες που έχει όσον αφορά την δική σας προεδρία και τις ε, δεσμεύσεις σας για την ε, θέμα της ε, συνδεσιμότητας στα πλαίσια της ανατολικής γειτονίας στην Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, γιατί η συνάδελφος μας μίλησε για τη Μολδαβία. Τώρα, για τη μεταφορά της πρεσβείας στην Ιεσουρουσαλία. Τι σχέση έχει αυτό με την μακροπρόθεσμη ε, πολιτική την οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη δύο κρατών συγχρόνων, Παλαιστίνης και Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο τελευταίος συνάδελφος. thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προτιμώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, άρα θα χρειαστεί να φορέσετε τα ακουστικά σας. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μια επιτυχημένη Προεδρία προϋποθέτει ότι οι προτεραιότητες της Προεδρίας σας θα λειτουργήσουν αυστηρά με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών και δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο θα πω ένα-δύο παραδείγματα για να ακούσω την άποψή σας κατά πόσο θα λειτουργήσετε με βάση αυτό το αυστηρό πλαίσιο και θα επικεντρωθώ στην Τουρκία. Μετά από πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω ίσως ένα-δύο χρόνια, ακούσαμε και τη φράση στρατηγικός εταίρος. Λοιπόν, γεγονότα. Η Τουρκία, για να κρυβολογούμε, η κυβέρνηση του Ερτογάν του ΑΚΠ δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνουν μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων το σεβασμό του rule of law στην Τουρκία, τον ελάχιστο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναγνώριση όλων των κρατών μελών περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλά άλλα. Θα προχωρήσετε σε αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων παραγνωρίζοντας όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Και το δεύτερο, Καθώς μιλάμε, στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε μία στρατηγική συνεργασία των εξής χωρών. Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και απέναντι Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Αίγυπτος, Ιορδανία. Απέναντι σε αυτή τη συνεργασία για σταθερότητα και ειρήνη έχουμε την κυβέρνηση του Ερτογάν. Μόλις σήμερα ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις, παράνομες ναύτεξ, εσείς τι θα προωθήσετε στην, περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Φυσικά προσδοκούμε ότι θα συνταχθείτε με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα οποία θέλουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ξεκινώντας από την Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο την Κύπρο. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Colleagues, may I σας ευχαριστήσω συνάδελφοι για τι ερωτήσει. σας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο 10 λεπτά, αλλά επιτρέψτε μου και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Μας είπατε ότι μία από τι προτεραιότητε σα θα είναι η ανατολική εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια τη προεδρία σα. Και ίσως θα μπορέσουμε να ερτάσουμε και την δεκατή επέτειο αυτής της εταιρικής σχέσης. Οι συνάδελφοι όμως τόνισαν την κατάσταση που επικρατεί στην Μολδαβία, που είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Συζητήσεις και εδώ και στην Ολομέλεια και η συντριπτική πλειοψηφία εκφράζει μεγάλες ανησυχίες για την ε, έλλειψη δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Η Προεδρία σας, λοιπόν, σκοπεύει να αναλάβει δράση για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Μολδαβία, κυρίως δεδομένου ότι έχουμε και βουλευτικές εκλογές την 21η Φεβρουαρίου. Thank you very much. I hope you will... Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μου επιτρέψετε Τα 7 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να... Α, δεν έχω 7, έχω 15. Είστε πολύ γενναιόδρος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν επιτρέψτε μου να απαντήσω στη δική σας ερώτηση που την έχω πρώτη. Θέλω να σας πω με απόλυτη σαφήνεια ποια είναι η θέση μας για τη Μολδαβία υποστηρίζουμε την προσέγγιση της ε, Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε καμία ειδική συμφωνία με κανέναν, στην Μολδαβία με κανένα πολιτική προσωπικότητα. Συνεργαζόμαστε με τα θεσμικά όργανα και Ο οργανισμός της περιφερειακής ανάπτυξης αφορά και την ανάπτυξη των πολιτών. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε σε σχέση με τις εκλογές, όπως είπατε κι εσείς ιδιαίτερος. Πριν από τρεις ημέρες, τέσσερις μέρες ίσως, ήμουν στο Κίτσινάου, συμμετείχα στην ε, ορτασμό της ημέρας της διπλωματίας και είχα συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών και το μήνυμά τους ήταν απόλυτα ξεκάθαρο. Υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα ξεπεραστεί. Είναι οι εκλογές. Θα πρέπει να γίνουν ε, με την ε, εποπτεία παρατηρητών από μας, από τον ΩΣΑ και να γίνουν απρόσκοπτα. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την κόκκινη γραμμή την οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουν ποτέ και το λέμε με απόλυτη σαφήνεια. Αυτά ήθελα να πω για αυτό το θέμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, επειδή έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις στα ρουμάνικα, επιτρέψτε μου να απαντήσω ρουμάνικα. Καλό είναι για εσάς, θα την καταλάβετε την απάντησή μου, οι άλλοι ίσως όχι. Ο κύριος Κριστιαν Πρέντα. Το θέμα της, επαν, της ε, ε Ένωση τη Ταϊβάν με την Κίνα. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στην 31η ε, Ιανουαρίου στο Βουκουρέστι. Με τη συμμετοχή όλων των Υπουργών Εξωτερικών και το θέμα αυτό θα συζητηθεί και η θέση όλων των κρατών μελών είναι μια θέση που θα υποστηρίξουν οι πάντες. Εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω το εξής. Πιστεύω ότι η επανένωση μέσω των διαπραγματεύσεων είναι η μόνη εναλλακτική λύση. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι πιστεύουν και οι συνάδελφοι το θέμα αυτό. Η μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ δεν είναι θέμα το μόνο που έγινε στην Ρουμανία μετά από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να μεταφέρει την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ είναι ότι κάναμε αξιολόγηση και ανάλυση του τι σημαίνει αυτή η κίνηση για την Ρουμανία. Εξετάσαμε τα υπέρ και τα κατά, αναλύσαμε την νομική βάση και τα στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι απόλυτα σαφείς οι αποφάσεις, άρα δεν έχουμε εμείς καμία απόφαση για την μεταφορά της πρεσβείας μας στην Ιερουσαλήμ, Μολδαβία. Είπαν ότι έχουν ε, μπλοκαριστεί οι διαπραγματεύσεις. Πολλές χώρες το έκαναν αυτό. Η δική μας η θέση ήταν αρκετά απλή. Κατά την άποψή μας, πριν από τις εκλογές δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε κανένα από τα κόμματα τα οποία είναι υποψήφια. Υποστηρίζουμε όσους θέλουν να κάνουν τις, δια... τις μεταρρυθμίσεις και Έχουμε σχέσεις με τα θεσμικά όργανα, όπως είπαμε, δεν έχουμε σχέσεις με άτομα προσωπικές. Τώρα, στο κύριο Κριστέα την ερώτηση. Προσδοκίες. Μετά από τις ε, εκλογές στη Μολδαβία. Εγώ ήμουν, όπως σας είπα, στην Μολδαβία πριν από τέσσερις μέρες. Συνάντησα τον Πρωθυπουργό και βεβαίως μίλησα εξ ονόματος Μίλησα, ε, συγγνώμη, με την πλειοψηφία και μίλησα και με εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Μετά από όλες τις συζητήσεις που είχα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή βασικά ένα τρίτο των ψήφων θα πάνε στους σοσιαλιστές, ένα τρίτο στους δημοκράτες και ένα τρίτο στην μη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση που έχει πολύ καλές προβλέψεις σύμφωνα με τις σφιγμομετρήσεις. Και εγώ είπα στην πλειοψηφία μην έχετε αγεφύρωτο χάσμα με την ε, μη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, μπορεί να τους χρειαστείτε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικά θέματα τα οποία θεωρούν σημαντικά διαφορετικά από αυτά τα οποία έχει η κυβέρνηση, αλλά τους είπα μην κόψετε εντελώς την επαφή. Δεν πρέπει να περιμένουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν οι εξελίξεις, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Όσον αφορά τη Σιγκαπούρη τώρα, η συνεργασία, η εμπορική με τις, με τις χώρες ΑΣΕΑΝ και τη Σιγκαπούρη. Όσον αφορά τις χώρες Ξέρουμε ότι έχουμε σχέσεις και διασυνδέσεις με την περιοχή αυτή και ένα τους κύριους μηχανισμούς τους οποίους χρησιμοποιούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε θέματα εκπαίδευσης για τους νέους. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητας, αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία διάσκεψη στο Βουκουρέστι μεταξύ Υπουργών Παιδείας των Ευρωπαϊκών Χωρών και εκείνων και μέσω και να οργανωθούμε με εκπροσώπους ε, ε, πανεπιστημίων και νέων και έτσι να συμμετάσχουμε στην ε, ε, ταχεία ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος στις χώρες αυτές. Και τώρα θα περάσω στα αγγλικά. Έχετε από 24 γλώσσες να διαλέξετε. Τι θέλετε μιλάτε. Ε, τότε θα έχω πρόβλημα. Τι μπορώ να πω. Έχει θετηθεί απόφαση από τη Βρετανική κοινωνία. Σεβόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγορία. Συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις μέσω του Μισελ Μπαρνιέ ε, με τις Βρετανικές αρχές. Και στο Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Δεκεμβρίου ε, εγκρίθηκε η συμφωνία περί αποχώρησης και η πολιτική διακήρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου αυτή την άποψη, αυτό μπορούμε να κάνουμε ως ε, ασκόντες στην Προεδρία, ως εκπεριτροπής Προεδρία τέλος πάντων του Συμβουλίου, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει παράταση της περίοδου αποχώρησης και στο μεταξύ προτείνει κάποιες τροπολογίες στο σχέδιο συμφωνίας ή στην πολιτική διακήρυξη, αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το πρόσφορο έδαφος ε, και τις διοργανωτικές προεργασίες ε, για να συναντηθούμε τις διάφορες χώρες και να επιτρέψουμε τη δημιουργία συνένεσης. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να συμφωνήσουν 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μεγάλη Βρετανία. Και θα σας έλεγα ε, ότι λυπάμαι πολύ για την απόφαση που λάβατε. Πραγματικά λυπούμε βαθύτατα για την απόφαση αυτή. Και μέλημα μα είναι να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όσο πιο κοντά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλεια, άμυνα, εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και σε πολλού άλλου τομεί. Ε, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια ισχυρή φωνή. Αν τώρα ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο φύγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός hard Brexit, έχουμε ε, το έγγραφο της στρατηγικής ε, εταιρική σχέσης που συνήψαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο το 2016 και αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση θα τη μετατρέψουμε σε νομική βάση για τη μελλοντική μας συνεργασία. Θα καλύπτει τις πολιτικές μας σχέσεις, την ασφάλεια και την άμυνα, τις οικονομικές σχέσεις, τις πολιτισμικές, την παιδεία, την καινοτομία και άλλους τομείς. Εμείς Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Πάντως, ως Προεδρία μπορούμε να προσφέρουμε τις διευκολύνσεις και να δημιουργήσουμε πρόσφορα έδαφος για να ανεβρεθεί το συντομότερο δυνατό συνένεση μεταξύ των συμβαλωμένων μέρων. Η κυρία Χάρμς μίλησε για την διαφθορά, για την Ουκρανία, Τουρκία, την παρέμβαση κτλ. Λυπάμαι, αλλά διαφωνούμε ως προς τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υποψήφιες χώρες ή τη σχέση με τα πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι η ύπαρξη ενός πυρήνα θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προσπάθειες να εφαρμοστούν αυτές οι θεμελιώδεις αξίες και σε άλλες χώρες, είτε είναι πλήρη μέλη είτε υποψήφιες χώρες, είναι από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της Ευρώπης στην δημοκρατική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών. Και αυτό ισχύει για σας, για μας και για την Τουρκία. Και θα απαντήσω στο πρόβλημα της Τουρκίας. Ειλικρινά σας λέω, περίπου ο μισός πληθυσμός της Τουρκίας, αν κοιτάξετε το δημοψήφισμα που έγινε, θα διαπιστώσετε ε, ότι ήταν οριακό το αποτέλεσμα, 50-50. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς, πώς μπορώ εγώ τι να πω, να απολαγούμε από τους Τούρκους και το μισό πληθυσμό που είναι υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το υπόλοιπο μισό της Τουρκίας προωθεί μια διαφορετική πολιτική. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και δεύτερον, στο μέτρο που έχουμε επαφέ με την Τουρκία, στο μέτρο που έχουν το καθεστώς υποψήφιες χώρες, θα έχουμε δυνατότητα κάποιες επιρροή. Αν κόψουμε τους δεσμούς, τέλος, τελεία και παύλα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ξέρω ότι διαφωνούμε, δεν θέλω να επιβάλλω τη γνώμη σε κανέναν. Εσείς αποφασίζετε, το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία και για τη Μολδαβία. Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και οι βλέψεις τους να γίνουν κράτη-μέλη είναι το σημαντικό, ο σημαντικότερος πυλώνας της δημοκρατικής μεταρρύθμισης στις χώρες αυτές, ακόμη και στη Ρουμανία. Αν Ούτε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Κανένα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει την τέλεια δημοκρατία. Ο διάλογο μα όμω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ω πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο διάλογο μια υποψήφια χώρα, ε, δίνει ε, ε ενάυσματα, υποστήριξη και ψυχώνει για την πορεία αυτή, τη δημοκρατική. Σας είπα λοιπόν για την Τουρκία τι πιστεύω. Ε, ο Υπουργό Κούκαν μας ζήτησε να σας καταπλήξουμε. Δεν μπορούμε να σας ξαφνιάσουμε και πολύ για να σας καταπλήξουμε. Πάντως αποφασίσαμε να οργανώσουμε σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στις 31 Ιανουαρίου ε, θα οργανώσουμε μια συζήτηση με συμμετοχή όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τα χαρτιά μας ανοιχτά και μάλιστα θα μας τιμήσει η παρουσία εκεί του Ντέβιτ Μακάλιστερ, γιατί ήδη είπατε ότι θα παραβρεθείτε και θα είναι σημαντική η ομιλία σας και η συμβολή σας στη διάσκεψη αυτή την υπουργική. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε, δεν ξαφνιάζει κανέναν, αλλά ε, ευελπιστώ τα αποτελέσματα να είναι για μερικούς από σας έκπληξη θετική. Υπουργέ, κύριε Πάσκου, κύριε Υπουργέ, είναι κανείς άπαξ υπουργός, είναι για πάντα υπουργός, γι' αυτό τον προσφωνώ έτσι. Κύριε Υπουργέ Πάσκου, θα ήθελα να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη είναι στόχος της Ρουμανίας και το λέω καθαρά και εξάστερα. Από τεχνική άποψη η Ρουμανία σέβεται πλήρως όλες τις προϋποθέσεις και πληρεί όλες τους όρους για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Ένα πρόβλημα μόνο υπάρχει. Το πρόβλημα είναι η ικανότητα των, πολιτών που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και χαμηλούς μισθούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώσουν όταν περάσουμε ε, στην Ευρωζώνη και θα το ευρώ. Γι' αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη και το, το χαμηλό εισόδημα, ώστε να μπορέσουν και οι πιο ε, χαμηλοί εισοδηματίε ε, να επιβιώσουν και μετά το πέρασμα στο ευρώ. Για να μην τους εξοντώσουμε με αυτή τη μετάβαση. Και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί η ιδέα Ευρω... Ευρώπης δύο ταχυτήτων ή μεταβλητής γεωμετρίας. Γι' αυτό και ένα βασικό μας μέλημα είναι να ζητήσουμε από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης, που έχουν το δικό τους νόμισμα. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα να προσκαλούνται στις συζητήσεις για δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, χωρίς φυσικά να αξιώνουμε να έχουμε και δικαίωμα ψήφου στη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να ενημερώμαστε και οι χώρε που δεν έχουν το ευρώ να ενημερώνονται για τη συζήτηση και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Ακόμη και εντό τη Ευρωζώνη. Για να μπορέσουμε κι εμεί να συνεχίσουμε το δρόμο μας προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Στόκες. Λέω ναι στη συνοχή ακριβώς, ακριβώς επειδή υπάρχουν προβλήματα και σε μας και σε άλλες χώρες. Η συνοχή και η σύγκληση είναι κατά τη γνώμη μας οι σημαντικότερες αξίες και θέλουμε να τις προωθήσουμε. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία της Προεδρίας να για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και στο ρουμανικό λαό τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ίσως αλλάξει η συμπεριφορά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσεις μας με την Ουγγαρία είναι εξαιρετικές. Και μπορώ να σας δώσω και ένα συγκεκριμένο επιχείρημα. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουγγαρία μας φέρνουν ως το δεύτερο μεγαλύτερο εταίρο τη Ουγγαρία. Πρώτη είναι η Γερμανία και δεύτερη η Ρουμανία στις εμπορικές συναλλαγές με την Ουγγαρία. Και ενισχύεται η θέση μας. Και έχουμε πολύ καλές εύρωστε οικονομικές σχέσεις. Και αυτό είναι προς το συμφέρον και των δύο λαών. Μπορεί να έχουμε κάποια διάσταση απόψεων ε, για μερικά θέματα, ιδιαίτερα μετά την εκατοστή επέτειο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αφήνουμε αυτά τα ζητήματα στους ιστορικούς να τα λύσουν. Πάντως, η προσωπική μου σχέση ε, ε, και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας και με τον Πρωθυπουργό, μπορεί να γελάσετε που θα σας το πω, αλλά είναι πολύ φιλική η σχέση μου και πιστεύω ότι θα βρούμε λύση. Κύριε Φρουτζουλίκα, μιλήσατε για τη διεύρυνση και πώς θα στηρίξουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της προσπάθειας σύγκληση και συνοχή. Για το Σέγγεν πληρούμε όλα τα κριτήρια, αλλά το πολιτικό ζήτημα μας ξεπερνάει. Επίσης έκανα ένα λάθος όταν μίλησα προηγουμένως για τις προτεραιότητες μας για τη σχέση με την ανατολική γειτονία. Έπρεπε να προσθέσω αμέσως και την νότια γειτονία. Γιατί έχουμε επίγνωση ότι όταν μιλούμε για τη μετανάστευση, για παράδειγμα, μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται το νότιο τμήμα της ε, Υπήρου. Από το Μαρόκο προς την Ισπανία οι ροές. Και θέλουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ Βορρά, Βαλτική θάλασσα, ανα, Ανατολάς, Ανατολής, εύξηνος πότος Μαύρη θάλασσα και νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεσόγειος θάλασσα. οδηγία για την, νομοποίηση, για την καταπολέμηση νομοποίηση όδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε, αυτή η οδηγία είναι σε φάση έγκριση στη Ρουμανία και ένα εκλεγή πρόεδρος ε, στη Μολδαβία και μεταφορά της ε, πρεσβείας. Ο κύριος Μαυρίδης ζήτησε για την προτεραιότητα που δίνουμε στην Τουρκία. Νομίζω τα απάντησε αυτά τα θέματα και ο κύριος Μακάλιστερ ε, έλαβε, ε, υπέβαλε τελευταία στην ερώτηση και έλαβε και μία απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριε Μελισκάνο. 20 πολύ εντατικά λεπτά προς το τέλος. Σας ευχαριστούμε για την επισκέψη στην Επιτροπή των Εξωτερικών. Ευχαριστώ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Μουλτσουμέσκ. Μουλτσουνορόκ. Α, Μουλνορόκ. Και καλή σας τύχη λοιπόν για, την, ε, για το εξάμεινο που ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Μελισσάνου, το χρειαζόμαστε. Αγαπητοί συναδελφοί, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα και γι' αυτό προτείνω να περάσουμε ευθύ αμέσω στο προσεχές θέμα που είναι το 32. So, colleagues, we come to item... Περνούμε στο 32, αγαπητοί συνάδελφοι της ημερήσιας διάταξης. Κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, παρακαλώ την κυρία Κανιέτε να λάβει το λόγο. Έχουμε προβλέψει 10 λεπτά βέβαια γιατί είχαμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τελευταία στιγμή χρειάστηκε αυτό το θέμα από τη χθεσινή ημερήσια διάταξη να έρθει στη σημερινή. Α εξηγήσει λοιπόν η κυρία Κανιέτα τη δική σα προσέγγιση, προσέγγιση για συνεργασία με του συνάδελφου των λοιπόν ομάδων και είμαι βέβαιο ότι η ομάδα μα θα ε, καταλήξει σε καλές συμβαστικές λύσεις για την έκθεση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αρχικά το θέμα αυτό όμω ήταν για σήμερα. Μετά το φέρανε μπροστά και τώρα ξαναγύρισε στη θέση του. Είναι τόσο σημαντικός εταίρος η Ρωσία δε, που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σε 10 λεπτά μόνο να τον συστήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα προσπαθήσω. 15 χρόνια διπλωματικών προσπαθειών έχω αφιερώσει για την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τη Ρωσία ως διπλωμάτης και ως υπουργό εξωτερικών. Ωστόσο από την ε, επίθεση κατά της Γεωργίας βλέπω ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει την πραγματικότητα ότι δηλαδή η Ρωσία από υπεύθυνο εταίρος διεθνούς κοινότητας μετατρέπεται σε ένα κράτος επικίνδυνο για τους γειτονές της. Και οι χειρότεροι εφιάλτες μου επιβεβαιώθηκαν το 2014 όταν προσήρτησε την Κρεμαία και ξεκίνησε έναν πόλεμο επιθετικό κατά της Ουκρανίας η Ρωσία. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι έχει πλέον έρθει η ώρα να σταματήσει η διπλωματική γλώσσα και πρέπει να κάνουμε αυτό που οφείλουμε, όπως άλλωστε το καταγράφω και στο σχέδιο εκθέσεως για την Ρωσία και τους γειτονικούς πληθυσμούς. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες στο σχέδιο εκθέσεως. Συνολικά έχουμε 375 τροπολογίες λάβει. Και βέβαια αυτό δεν μας ξαφνιάζει, καθώς πολλές από αυτές αναφέρονται στις ε, κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, κατά της Ρωσίας ε, λόγω των επικίνδυνων εγκληματικών δραστηριοτήτων και παραβίασης των όρων του διεθνούς κοινέου και δικαίου δεν επιτρέπεται να ανεχθούμε περισσότερο την παραβίαση του διεθνούς δικαίου κατά της Ουκρανίας ή άλλων χωρών. Πολλά είναι τα κράτη και οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει μια πιο αποφασιστική δράση με υποστήριξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι τροπολογίες βέβαια περισσότερο αναφέρονται σε μια νέα ε, νομοθεσία Μαγνίτσκι και πολιτική συμφωνία για παγκόσμιο ε, καθεστώς ε, κυρώσεων για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το πρότειναν ε, οι Ολλανδοί. Έχουμε αυτή τη στιγμή διακοπή της συμφωνίας, άρση της λειτουργίας της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριά σας λέει ότι πρέπει να σταματήσει η λειτουργία της, αλλά κάποιοι άλλοι προτείνουν την αντικατάστασή της από ένα νέο πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για οδήποτε πλαίσιο όσο η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει τμήμα της ε, Ουκρανίας και να προβαίνει σε πράξη επίθεση κατά των ευρωπαϊκών κρατών ευρύτερη. Η συνένεση μεταξύ μόνο ότι πρέπει να υλοποιηθεί η συμφωνία του Μίνσκ και να εμπλακεί πιο άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση της ε, σύγκρουσης. Μια ειρνευτική ε, δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον τόνο και επίση πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει χρόνος περιθώριο ή χρόνος ε, για να ή χώρος για να αναπτυχθούν διπλωματικές προσπάθειες. Αλλά έχουμε και τον αγωγό Nord Stream 2 και εγώ, η συγκεκριά αλλά και άλλοι συνάδελφοι, λένε ότι πρέπει να απευθύνει και πάλι έκλειστο το Κοινοβούλιο για να σταματήσει αυτό το έργο, καθώ δεν είναι ευθογραμμισμένο με την πολιτική για την ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι συνάδελφοι από την αριστερά του σώματο δεν συμμορίζονται την άποψη αυτή. Άρα, προσβλέπω σε πολύ καλέ συνεργασίε στην Επιτροπή, συνεργασία με του σκιώδει συγκητέ για την ενίσχυση των σχεσεών μας. Αύριο έχουμε την ε, πρώτη συνάντηση με πολλές συμβαστικές τροπολογίες που τις έχω ήδη συντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Sandra. That was excellent. That was... Εξαιρετικό κυρία Καρνιέτε, τόσο σύντομη και συγκεκριμένη. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και πίστερο χρόνο, αλλά θα μας πιέσει στο θέμα της Ινδίας. Έχω πέντε συναδέλφους. Μέχρι δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ. Κυρία Γιάκονσαρη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Συμβαστικέ τροπολογίε δεν έχουμε δει ακόμα. Θα πρέπει να τι συζητήσουμε βέβαια αύριο και λυπούμε πολύ που έρχεται τόσο καθυστερημένη η πρότασή σα. Μπα περιπτώσει, η ιδέα μου είναι η εξή η κύρια ιδέα, ότι είναι λυπηρό πω οι πολιτικέ σχέσει μεταξύ Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα εμεί να επαναλαμβάνουμε διαρκώ τα επιχειρήματά μα χωρί να βλέπουμε άνοιγμα ή κινητικότητα από την άλλη πλευρά. Λυπούμε πολύ λοιπόν. Η συγγήτρια πολύ η εισηγητρια πολυ σωστα στην παράγραφο υπαριθμών 4 επισημαίνει πω είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η αποκλιμάκωση των ε, εντάσεων και να επιδιωχθεί στη συνεργασία με τη Ρωσία η μείωση των κινδύνων για παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Μια σημαντική επίσημη πλατφόρμα είναι ο δικός μας ο διάκυβνο διάλογος, η ανταλλαγή επόψεων μεταξύ βουλευτών είναι εργαλείο ουσιώδες για την ελαχιστικοποίηση των κινδύνων ε, παρεξηγήσεων και παρερμηνεών Και γι' αυτό πρέπει και οι δύο πλευρές να αποδεθούν σε αυτή την προσπάθεια για την ε, απάλληψη των ε, προσκομμάτων, ώστε να ξεραρχίσει αυτός ο διάλογος και να φέρει αποτελέσματα. Είναι παράλογο να μην μπορούν να συναντούνται επισήμως οι πολιτικοί, ακόμα και όταν υπάρχουν, ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τεταμένες σχέσεις. Χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας που θα ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο, κυρίως σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και τομείς ε, κοινού συμφέροντος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Βεβαίως, όμως το ισχύον πλαίσιο πρέπει να παραμένει ενισχύ μέχρι ότου αντικατασταθεί από το προσεχές. Στην, προσεχή, στην παράγραφο 12 λοιπόν θεωρώ ότι σωστά ε, ζητεί υψηλό επίπεδο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και χωρών ε, με συμφωνίες σύνδεσης και ελεύθερο και ελεύθερο γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για την ενίσχυση και την ανάπτυξη διαλόγου υψηλού επίπεδου. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, πρέπει να εντείνουμε τις επαφές, τις διαπροσωπικές, να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση για ένα νέο Erasmus και ε, κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα βλέπω να μην το περιλαμβάνει η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης, δηλαδή οι συσχετισμοί μεταξύ κυβέρνηση της Ρωσίας, άκρας δεξιάς και εθνικιστικών κομμάτων ε, χωρών όπως για παραδείγμα η Ουγγαρία που απειλούν την δημοκρατία και τις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιακοτσάρη. Αγαπητή συναλφή, έχουμε ήδη μεγάλη καθυστέρηση. Παρακαλώ κάπως να μπορέσουμε να τηρήσουμε το πρόγραμμα. Μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά, μην προσπαθείτε να ε, εξαντλείτε το χρόνο. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και εκπροσωπώντας την κυρία Φωτίγκα, η οποία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να έρθει για λόγους ε, υγείας. Καλώς ορίζω την έκθεση Καρνιέτε. Η κυρία Καλιέτε γνωρίζει πολύ καλά τη Ρωσία, πολύ καλύτερα από πολλούς από εμά εδώ και διαγυγνώσει και την επεκτατική ε, πολιτική που αναπτύσσει στον Τόμπας και την Ουκρανία, στην ε, Συρία ακόμα, στις προσπάθειες υπονόμευσης αποσταθεροποίησης του Μαυροβουνίου, για, την οποία μάλιστα, για το οποίο μάλιστα είμαι εγώ, ε, συντάκτης της γνωμοδότησης, στην επίθεση κατά Ιων Σκρίπαλ, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη. Δεν φαίνεται να είναι λοιπόν φίλος μας ή να θέλει να υποστηρίξει τις αξίες και τις δημοκρατίες μας η Ρωσία. Η κυρία Φωτίγκα έχει ετοιμάσει λοιπόν τα σχόλιά τη μου στείλει να τα διαβάσω η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος εταίρος όσο συνεχίζει να συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο αυτό. Πρέπει να αναζητηθούν νέοι διάβλοι επικοινωνία να παραμένουν ανοιχτοί οι φυστάμενοι, αλλά βέβαια στο βαθμό του δυνατού. Ελπίζει σε καλή συνεργασία κατά την ε, επεξεργασία της εκθέσεως με την υιοθέτηση ενό κειμένου αντίστοιχου με αυτό του κυρίου Λάντσπεργκης όταν είχε εκείνο αναλάβει ο συζητητής την έκθεση και θέλει ιδιαίτερα να ε, αναφερθεί στην παράγραφο 10 με κόκκινη γραμμή για το ECR και ζητεί την ε, τροποποίηση του κειμένου έτσι ώστε να καλυφθούν ε, οι επιθυμίες και προτιμήσεις της ομάδας μας. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό το κείμενο και προσβλέψει συνεργασία με τη Σάντρα. Ευχαριστώ κύριε Σωστρεβίτσιος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω ε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Σάντρα Καλνιέτε για το σχέδιο έκθεσής της και προσβλέπω στην αυριανή συζήτηση των σχεδόν εισηγητών. Το σημείο αφετηρίας μας θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Γι' αυτό και ζητώ από τους ενδιαφερόμενους να μην έχουν ψευδεστήσεις ούτε ευσεβείς πόθους στην προσέγγιση των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Θα πρέπει η έκθεση να δράζεται σε μια αποτίμηση της πραγματικότητας και σε ρεαλισμό. Δεν πρόκειται εμείς να αλλάξουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει χαράξει την πορεία της και αυτή θα ακολουθήσει. Δεύτερον, γίναμε μάρτυρες ε, της διάρκειας εμπιστοσύνης ε, μεταξύ μου και των Ρώσων. Δεν υπάρχει καμία βούληση από ρωσικής πλευράς να διορθωθεί, να επουλωθεί αυτή η ε, απογοήτευση, αυτή η διάψευση της εμπιστοσύνης, ούτε υπάρχει πραγματική βούληση για ουσιαστικό διάλογο. Τρίτον, η Ρωσία επέλεξε την αυτοαπομόνωση και από πολλά ευρωπαϊκού θεσμού και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν είναι δικό μας λάθος η δική μας κακή εκτίμηση. Οπότε όταν μιλούμε για στρατηγική εταιρική σχέση, πραγματικά με ξεπερνά, δεν καταλαβαίνω. Τι είδου στρατηγική εταιρική σχέση θέλουμε. Η συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία είναι κάτι κενό, είναι κενό γράμμα και θα πρέπει να διακοπεί δεν έχει νόημα πια. Και τέλος, καμία ψευδέστηση για νέες ποιοτικέ σχέσεις με τη Ρωσία. Και μπορεί να θέλουμε κάποια συνεργασία, αλλά σε πολύ περιορισμένη βάση. Σε ό,τι αφορά την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, ούτε και αυτό το πολύ καταλαβαίνω. Τι ακριβώς εννοούμε. Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν είναι παρά Ρωσία είναι, μια ενισχυμένη Ρωσία. Είναι μια οικονομική και πολιτική σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Οπότε δεν μπορώ να... μην περιμένετε από μένα να καταλάβω κάτι που δεν καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι οι Ρώσοι. Είναι ένα ένα πρόσχημα για επέκταση ουσιαστικά. Γιατί λοιπόν εμπλακούμε σε κάτι που είναι ουσιαστικά το παιχνίδι της Ρωσίας και της επέκτασης της σφαίρας επιρροής της. Αυτό νομίζω είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση αυτής της, ε, αυτού του θέματος. Και ευχαριστώ και πάλι την κυρία Καλνέτε. Ευχαριστώ κυρία Στρεβίση Η Ρομπέκα Χάρμς. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, και τα συγχαρητήρια προς τη Σάντα Καλνέτε. Ε, αυτό το σχέδιο έκθεσης πολύ καλά περιγράφει τις προκλήσεις που μας έθεσε η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλο και περισσότερη στρατιωτική επέμβαση σε χώρες της ανατολικής μας γειτονίας, ακόμη και σε χώρες εταίρους μας. Από την άλλη πλευρά, η Σάντρα Καλνέτα περιέγραψε και κάποιους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με τη Ρωσία. Και επίσης τις απαντήσεις της σε αυτές τις αντιφάσεις προσδιορίζει ξεκάθαρα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και την αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα προτείνει και κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δημιουργηθεί καλύτερη κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ρώσων πολιτών και συμφωνώ με τις συστάσεις 15, 16 και όλα τα συναφή με την εμβάθυνση των ε, σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα διάβασα ότι στο μεταξύ ο Βλάντιμπερ Πούτιν έχει μεγαλύτερη υποστήριξη στη Σερβία από ότι στη Ρωσία, που είναι και η πατρίδα του. Οπότε φαντάζομαι ότι θα συνεχιστούν οι αλλαγές ε, στη Ρωσία και δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα πάρουν και ποια κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να εμποδίσουμε τις επαφές μας με τη Ρωσία, να τις κόψουμε. Ευχαριστώ, Ρεμπέκα, ο κύριος Φλέκερστεν και μετά ο κύριος Γιούρεκ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την καλή σας πρόταση. Πότε είναι μια διάκριση καλή. Όταν καταγράφει πιστά την πραγματικότητα, και το πράτετε εσείς αυτό, και όταν μας δίνει κάποια εργαλεία με τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και ίσως να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Και όντως το επιτυγχάνεται και αυτό, άλλωστε τα επισήμανε και η Ρεμπέκα ορισμένα από αυτά. Πλην όμως, θα μπορούσαμε να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι άλλο θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Δύο σημεία στα οποία δεν συμφωνώ τόσο το 21, όπου σας παρακαλώ ειλικρινά να αναλογιστείτε το εξής, ότι δεν είναι λάθος αυτό που λέγεται, αλλά υπάρχει άλλη πτυχή, γιατί το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι ο καλός, ο χειρότερος, ο κάκιστος, αλλά το πώς μπορούμε να απευθύνουμε μία έκκληση προς όλες τις πλευρές ώστε να σταματήσει αυτή η απαγόρευση των ταξιδιών για να ξανανοίξει ο διάλογος και το σημείο 13 με τον αγωγό Nord Stream 2 που ξέρω ότι δεν θα εξασφαλίσω συντριπτικές πλειοψηφίε ε, που θα με υποστηρίξουν αλλά πάλι πιστεύω ότι και η διαφοροποίηση στις πηγές έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μην κινδυνεύουμε να ακούμε απειλές ή να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κινδυνέψουμε από διακοπή σε προμήθειες από μεγάλους προμηθευτές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό παρακαλώ και το 2013 να το ξαναδείτε άλλωστε σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Νομίζω ότι έχει κάποια λογική. Στο 21 σου μπορέσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν και τελευταίος ο κύριος Γιώρακ. Σας ευχαριστώ. Η έκθεσή μας για τη Ρωσία, για την οποία ευχαριστώ την κυρία Καλνέτε, δεν μπορεί να παραβλέπει τον χαρακτήρα της σημερινής ε, Ρωσίας και του ιστορικούς της ε, δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση. Σχεδόν οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους αποτινάσοντας τη Σοβιετική κυριαρχία και η ασφάλειά μας εξαρτάται άμεσα από την διατήρηση αυτών των αλλαγών. Οι προηγούμενε εκθέσει και ψηφίσματα για τη Ρωσία αγνοούσαν το πρόβλημα τη παρακαταθήκη του πολσεβικισμού. Δεν θα ήθελα ε, η συγκεκριμένη έκθεση να κάνει το ίδιο λάθο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τη δημόσια λατρεία προ το Λένιν και άλλου ηγέτε πολσεβίκου, την απολογία του σοβιετικού υπεριαλισμού ή τη δικαιολόγηση του κομμουνισμού. Η καταδίκη του μπολσεβικισμού είναι προ το συμφέρον και τη Ρωσία, γιατί δεν νοείται ελευθερία χωρί χωρίς ε, ρήξη με το κομμουνιστικό παρελθόν και την κομμουνιστική παρακαταθήκη. Και ε, μην ξεχνούμε ότι η Ρωσία ήταν το πρώτο θύμα της θα καταθέσω και έκθεση που μιλάει για την επιτακτική ανάγκη ενίσχυση τη ανεξαρτησία των χωρών που την ανέκτησαν μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Και εννοώ για την τρέχουσα κατάσταση στη Λευκορωσία. Σήμερα η Ρωσία προσπαθεί να εξωθήσει τη Λευκορωσία να απαρνηθεί την εθνική τη κυριαρχία χρησιμοποιώντα την πίεση για τα ενεργειακά ζητήματα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αμελητή να προτείνει χρηματοοικονομική βοήθεια στη Ρωσία που θα αντισταθμίζει πιθανή διακοπή των ρωσικών επιδοτήσεων για την ενέργεια ενέργεια, καθώς και το Γενικό Σχέδιο Ενεργειακής ε, Ασφάλειας, ε, εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων. Η, η ανεξαρτησία της ε, Λευκορωσίας είναι θέμα όχι μόνο αίσθησης γεωπολιτικής ασφάλειας, γεωπολιτικής ασφάλειας για τις χώρες περιοχής, αλλά και της γεωπολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί είναι απαραίτητη εδώ η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε την ε, λευκορωσική ανεξαρτησία και θα πρέπει να το κάνουμε πάρα αυτά. Θα ήθελα αυτή η τροπολογία να ληφθεί υπόψη στο ψηφισμά μας. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Δεν βλέπω άλλον κανένα. Οπότε Σάντρα, έχεις να προσθέσεις κάτι. Αύριο, αν κατάλαβα καλά, θα συναντήσει τους και ηγετές για να εξετάσετε τις συμβαστικές τροπολογίες. Ναι, είχε προβλεφθεί για τις 10 η αυριανή μας συνεδρίαση, αλλά μια και συνεχίζεται η σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών, μόνο οι πρώτες 15 έχουν ετοιμαστεί, Φαντάζομαι γύρω στις 8 θα μπορέσουμε να στείλουμε και τις υπόλοιπες, τις πρώτες 15 τις στείλαμε, αλλά ίσως χρειαστούμε και δεύτερη συνεδρίαση των, των σχεδόν εισηγητών για την επόμενη εβδομάδα. Πάντως αύριο στις 10 ανακρατήσουμε την πρώτη μας συνεδρίαση και πρώτη συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, που έκαναν προτάσεις για την έκθεσή μου και περιμένω με ανυπομονησία την ε, επικοδομητική συνεργασία με τους και ηγητές. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Μας έμεινε μόνο μισή ώρα για τις 5.30 έχουμε την κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Ανάπτυξη. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε. Καλό τον Τζέφρι να έρθει να καθίσει δίπλα μου. Και τον κύριο Βίγκαντ. Πού είναι ο κύριος Βίγκαντ? Α, εκεί είσαστε, εκεί πίσω. Herzlich willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Wir müssen das ein bisschen abkürzen. So. So, colleagues, I welcome... Να, αδελφέ, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ιγύριο Βίγκαν που θα μας παρουσιάσει τη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας που κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, να καλωσορίσω του συναδέλφου εδώ και δίνω αμέσως τον κύριο Βίγκαν λόγο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Με καλείτε δηλαδή να μιλήσω πολύ γρήγορα. Θα προσπαθήσω να εστιάσω στα κύρια σημεία και να σας εξηγήσω ποια είναι η πρόταση και η ανακοίνωση της Επιτροπής και της ε, είπα της εκπροσώπου που παρουσιάστηκε τον ε, Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, μετά από τρεις εβδομάδες, εγκρίθηκε και από όλο το Συμβούλιο. Ήρθαμε από πριν από το, το πριν από 10 μέρες, περάσαμε κάποιες μέρες ε, με τους ε, εκπροσώπους ε, στο Συνδία, στον Ιδελχή και άλλους εκπροσώπους άλλων κρατών της περιοχής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Ινδίας έκανε και μία ανακοίνωση στον τύπο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών για να καλωσορίσει αυτή την ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στα πλαίσια των εξωτερικών ε, σχέσεων της Ινδίας. Με άλλα λόγια δηλαδή πρέπει να πω ότι έχουμε μια παρεμφερή προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο θα εμβαθύνουμε και θα ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας. Διότι Πριν από 14 χρόνια είχαν γίνει οι πρώτες προτάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ινδίας για συνεργασία και θα ήθελα τώρα εδώ να ζητήσω από τις ε, εμπλεκόμενες κοινωνίες ένθεν και ένθεν να προσπαθήσουν να ενισχύσουν αυτή την συνεργασία. Πιστεύω ότι τα θέματα ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι από τα κύρια θέματα, καθώς και οι προκλήσεις στον κόσμο σήμερα. Όλα αυτά θα γίνουν, πρέπει να γίνουν μέσω συνεργειών και μεγαλύτερης ε, σύγκλησης και συνοχής μεταξύ ημών και ημών, κάτι το οποίο δεν ήταν πάντα χαρακτηριστικό των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Ινδία. Θέλουμε λοιπόν να επωφεληθούμε από αυτή την δυναμικότητα που παρουσιάζει αυτή η εταιρική σχέση, ώστε να υπάρξει αηφόρος ε, εξυγχρονισμός της Ινδίας, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για την Ινδία και για τις πόλεις και για την οικονομική της διάθεση. Επίσης θα πρέπει να ε, μπορέσει με την πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ διεθνών οργανώσεων και Ινδίας να βελτιωθεί και ε, η κοινωνία αυτή που είναι η δεύτερη πιο δημοκρατική μεγάλη χώρα και σημαντική για την ε, σε εμπορικές σχέσεις και την οικονομία της αγοράς σύνομα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε πώς τα σημερινά θέματα που μας απασχολούν και μας προκαλούν, η κλιματική αλλαγή, τα θέματα ασφαλείας, να τα λύσουμε από κοινού και να τα προχωρήσουμε. Η αντιπροσωπεία μας με πολλές φορές τόνισε πώς σημαντικά είναι αυτά τα θέματα στην Ινδία. Η Ινδία βεβαίως είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από γεωπολιτικής πλευράς είναι εταίρος σημαντικός δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Σήμερα η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία μετά τις χώρες της ΑΣΕΑΝ. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ευημερία και να εστιαστούμε περισσότερο στον συγχρονισμό της κοινωνίας, τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Είμαστε λοιπόν εξαιτίας, τη... συγγνώμη, χάρη στην τεχνογνωσία την οποία έχουμε και τις ε, τεχνικές μας γνώσεις ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για την Ινδία και σε διάφορα θέματα, κυρίως ενεργειακά, είμαστε αυτοί που έχουν την πραγματική πραγματογνωσύνη. Έχουμε νέες δυνατότητες εμπορικές και από τις δύο πλευρές και βεβαίως προ... θέλουμε να προωθήσουμε ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ινδία είναι πραγματικά αξιοσημείωτες. 6.000 εταιρείες ε, δίδουν δουλειά σε 6 εκατομμύρια Ινδούς. Και οι επενδύσεις ε, είναι της τάξης των 73 και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ινδία να αναπτυχθεί. Επίσης είναι κάτι, κάτι που πρέπει να διευκολύνουμε είναι η εύκολη μετακίνηση φοιτητών, ερευνητών, κέντρων καινοτομία κτλ. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ε, στρατηγική διασυνδεσιμότητας, πράγμα το οποίο συζητήθηκε εδώ και προηγουμένως. Η στρατηγική διασυνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα πρέπει σε να αναπτυχθεί με εταιρικέ σχέσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα που βρίσκεται πιο κοντά στην Ευρώπη από τις άλλες. Δεν θέλουμε εδώ να εξετάσουμε μόνο μία διμερή ε, σχέση, αλλά μία σχέση η οποία θα αποτελεί απόκριση στις προκλήσεις που τίθενται στην περιοχή εκείνη. Το θέμα της ε, ε, συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας είναι κάτι το πολύ σημαντικό έχουμε αρχίσει να κάνουμε σημαντικό διάλογο για θέματα που μας αφορούν όπως η μη διάδοση των ε, ε, όπλων μαζικής καταστροφής, θέματα ασφάλειας των, ε, για την ακτοφυλακή της Ινδίας και άλλα θέματα. Την επόμενη εβδομάδα το ότι θα φτάσει το πλοίο ε, Κασά, το γαλλικό, είναι κάτι το οποίο θα εντείνει τη συνεργασία. Συμπερασματικά πρέπει να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να μπορέσουν ε, να γίνουν σεβαστοί όλοι οι κανόνες που πρέπει να διέπουν ε, τις ε, χώρες μας και να λάβουμε υπόψη ότι στην σημερινή κατάσταση των πραγμάτων θα πρέπει για την κλιματική αλλαγή και για άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα από κοινού στα πλαίσια της παγκόσμιας τάξης. Και με τον τρόπο αυτό θα αποδείξουμε ότι υπάρχει συνοχή. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας, δεδομένου ότι με την εργασία αυτή επιτελέσαμε αυτό το οποίο ζητήσατε εσείς το 2017. Όταν ζητήσατε να υιοθετηθεί στη σχέση μας με την Ινδία μία προσέγγιση συνεκτική. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Βίγκαν για την παρουσίαση. Και παρακαλώ τον κύριο Βανόρντι να λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενθαρρυντικά τόσο ακόμα αυτή η νέα θετική προσέγγιση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και καλωσορίζω και την αποδοχή από την Ινδική κυβέρνηση των νέων αυτών δράσεων. Η Ινδία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει πολύ από την εγκαθίδρυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2004 πρέπει να πούμε. Θα θυμάστε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη τη χρονιά προχώρησε στη διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη. Και ήταν ήδη τότε 12η σε ταξινόμηση ΑΕΠ η Ινδία. Ενώ τώρα είναι έκτη. Αφού είναι μετά την ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα γίνει, αναμένεται, να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο στο εγγύς ε, μέλλον. Ξέρετε, Πρόεδρε, ότι είμαι επικεφαλή ε, τη αντιπροσωπεία ε, για τη σχέση με την Ινδία και από τότε που ανέλαβα έχουμε ιδιαίτερη έμφαση δώσει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ινδία και κρατών μελών και βελτίωση τη γνώση για την Ινδία και την πολιτική ζωή της στο Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θα σας κάνω ε, εκτενή αναφορά στις δραστηριότητες μας τα τελευταία, τελευταία πενταετία. Ήταν όμως πολλές και ποικίλε. Η οικοδόμηση όμως αυτών των θετικών σχέσεων θέλω να πω δεν μπορούσε παρά να στηριχθεί ή να έχει προκύψει κατόπιν μιας ευνοϊκής ε, Αμέλεια τη ευρωπαϊκή Ένωση θα την αποκαλέσω έτσι και αφορά αυτή όχι μόνο την Ινδία αλλά και άλλε χώρε ε, που λίγο έχουν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο ενδιαφέρον έχουν δει δηλαδή πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Βίγκαν ε, αυτό καταγράφεται και στο ε, ανακοινωθέν. φαίνεται να υπάρχει όμως μία πρόοδος ως προς τη σημασία των, της συμφωνίας για τις συνολικές οικονομικές σχέσεις. Είναι σελίδα 7 λέγεται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το εμπόριο, η επενδύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας και να προχωρήσουμε σε ολιστικές και γενικές εταιρικέ σχέσεις. Τα λόγια αυτά είναι θετικά με μεν, αλλά δεν θεωρώ ότι αποτελούν ουσιαστική πρόοδο σε σχέση με τη διατύπωση του ανακοινοθέντος του Οκτωβρίου 2017 στη Συνοδοκορυφής 10 σελίδες, 53 παράγραφοι ήταν το ανακοινωθέν εκείνο και κατέγραφαν τις σχέσεις με μία μόνο αναφορά στην ε, Συμφωνία εταιρική Σχέσης ε, Ελεύθερων Συναλλαγών. Ε, πολύ λίγα λόγια λοιπόν για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ε, συμφωνίες εμπορίου που 12 χρόνια τώρα επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ινδία, η ΣΥΤΑΤ του Καναδά, η ΣΥΤΑ με τον ε, Καναδά. Χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί. βεβαίω αν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση και βεβαίως ότι υφίσταται κάτι τέτοιο στη σχέση μεταξύ Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίε. Ξέρουμε ποια είναι τα διαφιλονικούμενα ζητήματα. Πρέπει να πω ότι είναι ευπρόσδεκτη η τομεακή συνεργασία που περιγράψατε σε διάφορους τομείς. Οι σχέσεις μας ξεπερνούν τις οικονομικές αυστηρά σχέσεις. Έχουμε πολλά, κοινά συμφέροντα, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το είπατε και εσείς, ε, ε, καθαρή ενέργεια, κλιματική αλλαγή, καθαρές θάλασσες. και ως ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την ότι για μια χώρα που η οικονομία της είναι η, μεγαλύτερη, η έκτη μεγαλύτερη του κόσμου και που ταχύτατα μετατρέπεται στην μεγαλύτερη σε χώρα, τέταρτη σε στρατιωτική δύναμη, οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε δεν έχει δεχθεί την αναγνώριση και τη σημασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα τι άξιζε. Ενώ υπάρχουν τόσοι τομείς στου οποίου δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και ελπίζω και αυτή η ευκαιρία να αναγνωριστεί πλέον, να μην χαθεί. Πολλοί είναι οι τομείς στου οποίου έχουμε ξεκινήσει συνεργασία, πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Και ελπίζω πια να αποσταλεί και να γίνει δεκτό και το μήνυμα ότι άλλαξαν οι καιροί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Jeffrey Ευχαριστώ κύριε Βανόρντεν. Μερικά λεπτά μας μένουν ακόμα για τις ανταλλαγές απόψεων. Πρέντα, Τάνακ, Λόχπιλερ. Ξέχασα κανέναν. Μπασίρ. Ωραία. Με τον κύριο Πρέντα λοιπόν ξεκινάμε κλείνοντας τον κατάλογο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 2017 ανέλαβα εισηγητής εκ μέρου του Κοινοβουλίου για τις ε, πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ένωση και Ινδία. Ιδιαίτερη έφαση λοιπόν είχα δώσει στην ε, στρατηγική ένωση, στρατηγική σχέση με την ε, Ινδία. Χαίρομαι λοιπόν που πλέον θεσπίζουμε, ορίζουμε προτεραιότητες για μια πραγματικά, μια γνήσια στρατηγική εταιρική σχέση Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να υιοθετήσουν την ανακοίνωση επιτροπή. Χαίρομαι γιατί αυτό αποτελεί ένα σαφέ μήνυμα προ τι αρχέ τη Ινδία. Επιβεβαιώνει δε την προσήλωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόοδο στι σχέσει. Βεβαίω πρέπει πλέον, ε, αφού εντοπίστηκαν οι προτεραιότητε, να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Και θέλω, κύριε Βίγκα, να μου, να μου περιγράψετε τα προσεχή βήματα. 11-12 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε, αναμένεται η επίσκεψη του κύριου Γκοκάλα, Υφυπουργού Εξωτερικών ε, για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, ε, στις Βρυξέλλες, τι περιμένετε, τι πρόοδο διαβλέπετε και επίσης ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ινδία. Πώς διαγράφεται μια τέτοια προοπτική, γιατί πολλές πληροφορίες δεν έχουμε από τα δύο έγγραφα. Μόνο από τα ανακοινωθέν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου βλέπω μια αμνία. Ε, Μουτσομέσκ, Κρίστιαν Τσάλ Στάνακ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν από 20 χρόνια, 20 χρόνια είμαι στο Κοινοβούλιο, το 1999, μαζί με τον Τζέφρι Βαν Όρντεν, θεσπίσαμε την ομάδα Φίλη της Ινδίας, που διελήθη όταν δημιουργήθηκε η αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Ινδία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το επίσημο όργανο αυτό βέβαια σήμαινα, σήμανε και την αναγνώριση ως περιφερειακής δύναμης της Ινδίας, ε, που είναι μία από τις BRICS, πέμπτη σύντομα οικονομικά δύναμη, θα προηγηθεί δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, με μεγάλη ιστορική σημασία στη σχέση της με την Ευρώπη, όπως άλλωστε και η Κίνα από τον 17ο, 18ο αιώνα. Ε, Κοινέ λοιπόν δημοκρατικές αξίες, σεβασμός του κράτου, κράτους δικαίου, πολύτιμος ε, τέρος εμπορικός, σημαντικός και για τα θέματα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατίας, γιατί μπορούμε σε στενή συνεργασία να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πυρηνική δύναμη. Οφείλω να πω ότι θα ήθελα να είναι και μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας ως τέτοια. Ε, αποστέλει τακτικά ειρηνευτικές αποστολές. Σημαντική και στη σχέση με την Αυστραλία και την Ισλανδία. Και εκεί θεωρώ ότι θα είναι λυπηρό ότι με την αποχώρηση του Ρωμανού Βασιλείου από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγκαστεί να περιοριστεί μόνο σε διμερείς σχέσεις με την Ινδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν ε, εκείνο από ό,τι φαίνεται και είναι παράδοξο αυτό ε, είχε τις αντιρρήσεις του στην πρόοδο στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τώρα στην απαλλαγή από τη θεώρηση διαβατηρίων που προβλεπόταν. Ε, εν πάση λοιπόν, με το Brexit ίσως θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει αυτή τη φιλόδοξη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τα σημαντικά πλέον εκτήματα και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο εταίρων. Ευχαριστούμε, Τσάρς. Κυρία Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Βίγκαντ που μας παρουσίασε τη στρατηγική για τη σχέση με την Ινδία. Σε όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα να, αυξήσουμε, να ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν κάποια σχέδια για συνεργασία με την Ινδία προκειμένου να ενισχυθεί η πολυμέρεια και ενδεχομένως ε, να προβληθούν κάποια θέματα για ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενενέβη ή στο Ηνωμένο Έθνη βλέπουμε και στα ψηφίσματα ότι έχουμε πολύ καλές νομοθεσίες και στην ε, Ινδία για την πρόθεση και προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα στην πράξη έχουμε βία κατά των γυναικών, ε, πρόσφατες ε, συλλήψεις ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πράξη λοιπόν δεν ανταποκρίνεται στη θεωρία που προβλέπει καλή κατοχήρωση των ανθρωπίνων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα λαμβάνεται αυτά υπόψη στη στρατηγική. Επίσης, μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να συζητήσουμε κάποια θέματα συγκρούσεων ε, στην ευρύτερη περιοχή. Μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα γίνουν κοινέ προσπάθειες για να εξεταστεί η κατάσταση στη Σρι για παράδειγμα. Ε, για παράδειγμα, δεν ε, έχει εξεταστεί το θέμα των, της διάπρεξης εγκλημάτων πολέμου. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα εκεί. Ο κύριος Μπασίρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ώρα περνάει γι' αυτό και δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι πολύ σωστά εκτιμούμε τη παγκόσμια δημόσια τάξη που θα εδράζεται σε κανόνες και το Ηνωμένα Έθνη που είναι ετοιματίσει. Έχουν περάσει πολλά ψηφίσματα στα Ηνωμένα Έθνη για το Κασμίρ που δεν έχουν εφαρμοστεί και πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται στο Κασμίρ. Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε στην Ινδία τις υποχρεώσεις που φέρει να τηρήσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να ε, διαθετήσει αυτή τη διαμάχη ώστε να μην έχει 700.000 ε, ε, στρατιωτικούς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κασμίρ. και από το 1989 περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ υπάρχει ατιμορρησία, ασυλία για τις ένομιλες δυνάμεις της Ινδίας ε, που βρίσκονται στο Κασμίρ. Κάτι που παραβιάζει κατάφορα τις δικές μας αξίες. Αν λοιπόν η Ινδία είναι μια οικονομική δύναμη, τότε δεν θα πρέπει να τη δεχτούμε μόνο επειδή είναι τόσο επιτυχής. Θα πρέπει να ζητήσουμε ε, να εστερνίζεται και τις υπόλοιπες ε, θεμελιώδεις αξίες μας. Σας ευχαριστούμε. Ποιος θα ήθελε πρώτο το λόγο, Τζέφρι εσύ, πρώτα εσύ και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίγκαντ. Πολύ σύντομα. Ο κύριος Μπασίρ επισήμανε αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα του Κασμίρ. Το Κασμίρ είναι μια πολιτεία της Ινδίας, είναι ένα κράτη της Ινδίας και ένα τμήμα του Κασμίρ ε, βρίσκεται υπό πακιστανική κατοχή αυτή τη στιγμή. Το Κασμίρ, το Γκυλγκίτ και το Μπαλτουστάν. Και ε, εξετάσετε εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, βλέπετε πόσο επικριτικές είναι για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το τμήμα του Κασμίρ, όπου ο πληθυσμό υπόκειται σε τεράστιες κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επίσης είναι και πλατφόρμα ε, ε τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της Ινδίας. Είναι φαλτήριο των τρομοκρατών. Και Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και νομίζω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον μια ειρηνική συνύπαρξη Ινδίας και Πακιστάν και μια διαθέτηση των διαφορών τους ώστε να δημιουργηθούν οικονομική δεσμοί και δεσμοί μεταξύ των κοινοτήτων. Και υπάρχει αρκετή προθυμία και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν θα βοηθήσει μια μεροληπτική μόνο θεώρηση της κατάστασης που μερικές φορές παρουσιάζεται σε φόρα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε, για την υποστήριξη και για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, νομίζω ότι είναι αναφίβολο ότι υπάρχει ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαπραγμάτευση μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία. Και μάλιστα στα συμβούλια του συμπεράσματο αναφέρεται η σταθερή δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ μια ε, φιλόδοξη, αμοιβαίω επωφελή και σφαιρική συμφωνία για το εμπόριο και τι επενδύσει με κανόνε που θα συνάδουν και με την αηφόρο ανάπτυξη. Και το νέο πλαίσιο προστασία επενδυτών θα προσελκύσει περισσότερε ευρωπαϊκέ επενδύσει στην Ινδία. Οπότε η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά και οι εργόντες προσπάθειες του επικεφαλής διαπραγμάτευσης είναι να βρεθούν κοινοί ορισμοί για το τι εστί σφαιρική, περιεκτική, φιλόδοξη και αμοιβαίως επωφελής και οικονομικά βιώσιμη συμφωνία. και δεν έχουν λυθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες και ποια είναι η εμβέλεια αυτής της συμφωνίας και ποιο το πεδίο εφαρμογή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο συμφωνία χωρίς κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης ή κεφάλαιο για το εμπόριο και τη δημόσια ανάπτυξη, για τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν αναφέρεται τίποτα για τις ε, δημόσιες συμβάσεις ή αν δεν έχουμε εκτενή κάλυψη των εμπορικών αγαθών ή των υπηρεσιών. Οπότε υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν εκκρεμότητες και θα πρέπει να συνεχίσουμε και να βαθύνουμε τις προσπάθειές μας. Πάντως υπάρχει βούληση από ειδική πλευράς για μεγαλύτερη ευέθυνση, για καλύτερο προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογή. Μπορεί να μην είναι τελικά η ευέλεια τόσο μεγάλη όσο άλλες προηγμένες ε, εμπορικές συμφωνίες, αλλά θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ, ώστε να μην είναι μόνο ε, περιορισμένη στον ΠΟΕ, αλλά πιο ευρεία. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Πρέτα, όντως ε, ο υπέξ της Ινδίας θα έρθει σε δύο εβδομάδες εδώ και θα έχουμε πολλές συνομιλίες και επαφές και με το Γενικό Γραμματέα και προβλέπονται πολλές εκδηλώσεις και διασκέψεις και θα έχουμε ε, ειδικευμένε διαβουλεύσεις και για θέματα ασφάλειας και για οικονομικά θέματα και αργότερα μες στο έτος θα γίνει και διάσκεψη κορυφής μετά το πέρας των ευρωεκλογών και μετά και τις συνδικές εκλογές για να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ισοαμιλητές μας και από τις δύο πλευρές. Πάντως, Υπάρχει πολιτική συμφωνία μεταξύ των πρόεδρων του και Γιούγκερ και τον πρωθυπουργό Μόντι όταν πρόσφατα συναντήθηκα στον Πόενο Άιρες στη διάσκεψη κορυφής του G20. Και η ανάγκη να είμαστε προορατικοί εδώ και να φροντίσουμε να προωθήσουμε τις προτεραιότητες μας και να μην μείνουν όλα αυτά σε επίπεδο αγαθών προθέσεων, όπως μας είπε ο κύριος Στάνοκ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι καθήκον μας να τα προωθήσουμε. Και έχουμε πολύ στενότερη συνεργασία, όπως θα ήθελα να πω στην κυρία Λοχπίλερ, γιατί έχουμε κάποιες ε, αλλοκαλυπτόμενες γειτονίες, Μέση Ανατολή, Αφρική, και συνεργαζόμαστε με την ίδια και στις περιοχές αυτές, αλλά ε, θα συνεργαστούμε και για κάποιες καταστάσεις στην Ινδική γειτονία και το έχουμε κάνει με πολύ αγαστή συνεργασία. Όταν πρόσφατα είχαμε δυσκολίες σε χώρες που αναφέρατε, στις Μαλδίβες, στη Σρι Λάγκα, γιατί μας ενδιαφέρει η συνταγματική τάξη, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου να παραμείνουν στις χώρες αυτές. Επίσης, μας ενδιαφέρει καλύτερη συνεργασία με την Ινδία και την κατάσταση σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές ή η Μιανμάρ. Τέλος, να απαντήσω στην ερώτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώ και το Κασμίρ ειδικώ. Επιδιώκουμε στενότερες ε, επαφές και συνεργασία με την Ινδία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό φαίνεται και στα έγγραφα του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η Ινδία συμμετέχει και πάλι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και προτείνουμε ημερομηνία για τον επόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός εταίρος. Η Ινδία έχει α, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχει μείνει και τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να επαναληφθεί. Πάντως παρακολουθούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία και στηρίζουμε, τους στηρίζουμε με ευαισθητοποίηση, με χρηματοοικονομική υποστήριξη και άλλα μέσα που μας δίνει ο Μηχανισμός Γειτονίας Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, προσπαθούμε να αποφύγουμε διακρίσεις λόγω κάστας, φύλου και βία. Και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χειραφέτηση των γυναικών. Ε, σε ό,τι αφορά το Κασμίρ είναι σαφή η θέση μας. Ανθαρρύνουμε και την Ινδία και το Πακιστάν να αναζητήσουν μια βιώσιμη λύση προκειμένου να διευθετηθεί η κατάσταση στο Κασμίρ με την ανάμειξη στο μέτρο του δυνατού του ίδιου του λαού του Κασμίρ. Και είναι ευθύνη και των δύο χωρών να διατηρήσουν ειρηνικέ σχέσει και να βρεθεί λύση στις διαφορές τους. Θεωρούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να διελευκανθούν, να διερευνηθούν άμεσα και με διαφάνεια με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις και εκτιμούμε το γεγονός ότι η Ινδική κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι, ε, δέχεται πρέσβης από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπει μετάβασή του στο Κασμίρ και συνεργαζόμαστε με την Ινδία και το Πακιστάν για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τις τρομοκρατικές απειλές πάσης φύσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκαντ. Άλλα σχόλια από πλευρά σας. Όχι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βίγκαντ που ήρθατε. για τη συνεργασία αυτή, για τη συνάντηση με την ΑΦΕΤ. Το επόμενο και τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το υπαριθμό 34. Και το λέω καθώς κάποιοι από μας είναι εδώ στην αίθουσα από τις 9 το πρωί. Είμαστε εδώ στην αίθουσα από τις 9 το πρωί. Αλλά είμαστε έτοιμοι, ορεξάτη, για τη συνεδρίαση την κοινή με τους συναδέλφους της ΔΕΒΕ που μπαίνουν σιγά σιγά.